Ready? So, my dear colleagues, chers amis, installez... Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Παρακαλώ καθίστε. Voilà, prenez place pour cette 60 για την 74η συνεδρία Συμμεκτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μας. Θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας με μια πολιτική συζήτηση. Υψηλού επίπεδου, γιατί βλέπετε ότι έχουμε στο βήμα Έχετε καθίσει όλοι. Ωραία. Ε, In Turkish? 25 for Turkish. Για τα τουρκικά στο κανάλι 25. 25 επαναλαμβάνω. So, bonjour à tous. Καλημέρα σε όλους. Άρχεται η 74η συνεδρίαση της κοινή 74η ε, συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μας με πολιτικό διάλογο υψηλού επίπεδου. Βλέπετε ότι είναι εδώ ο Υπουργός της Τουρκίας για τα ε, ευρωπαϊκά θέματα. Ε, τον γνωρίζετε. Έχουμε τον επίτροπό μας, ε, τον κύριο Φούλε, που θα μας πει ορισμένα πράγματα και για τη σχέση, για την κατάσταση των σχέσεων μας με την Τουρκία, αλλά και για να απαντήσει και στα ερωτήματά σας. Ο Έλληνας πρέσβης που είναι εδώ και ο οποίος θα λάβει το λόγο εκ μέρους της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου. Και θα θυμάστε ότι η τελευταία μας συνεδρίαση ήταν το Δεκέμβριο του 2013. Από τότε είχαμε την ε, ευκαιρία μέσω της ε, κοινοβουλευτικής μας ε, έκθεσης μπορέσαμε να εκφέρουμε άποψη σε σχέση με την κατάσταση στην Τουρκία αλλά και, με τις, και στις σχέσεις μας και των, των σχέσεών μας με την Τουρκία. Είναι εδώ η ε, συνάδελφος ε, Ρία Όμεν Ρόιτεν, η οποία μετά τους ε, προσκεκλημένους μας θα λάβει και εκείνη το λόγο για να μας υπενθυμίσει τις προτεραιότητες και τους βασικούς άξονες της εργασίας της στο πλαίσιο της έκθεσης για την Τουρκία. Υπάρχουν επίσης και κάποια γεγονότα στην επικαιρότητα, οι εκλογές στην Τουρκία, στη Γαλλία και τοπικές εκλογές ε, των οποίων ε, προηγήθηκαν ε, πολλές, ομάδες, πολλές εβδομάδες και πολλοί μήνες περίπλοκων διαδικασιών και ταχύτατων αλλαγών στην Τουρκία για τις οποίες θα μιλήσουμε. Έχουμε ειδικό θέμα ε, όσον αφορά τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία. Θα συζητήσουμε για τα πάντα, για το ε, ε, για το Συμβούλιο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο στην Τουρκία, όπως επίσης και για την νομοθεσία για το ίντερνετ. Ούτως ή άλλως είχαμε ακούσει από τον αρμόδιο υπουργό, πρωθυπουργό για τα θέματα αυτά και βέβαια θα ακούσουμε ορισμένα πράγματα και για τις ε, κοινωνικές, για την κοινωνική κατάσταση ε, στην Τουρκία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα γεγονότα, τα οποία σχολιάζονται συχνά ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Με τον ε, κύριο Ντεμίρ ε, θα ε, συζητήσουμε για τη συνέχεια των εργασιών μας μετά για να μην αργήσουμε και θα προτιμούσα να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους γιατί θα πρέπει να φύγουν οι προσκεκλημένοι μας σύντομα και ο Επίτροπος αλλά και ε, ο πρέσβης ο κύριος Σωτηρόπουλος. Θα δώσω λοιπόν ε, στους προσκεκλημένους μας πρώτα το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο σε εσά ε, για ερωτήσεις, αρχίζοντας βέβαια με την κυρία Όμεν Να δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στον κύριο Φούλε. Αν μου επιτρέψετε θα πω κι εγώ ένα καλημέρα στα τουρκικά. Θα ήθελα και εγώ να πω καλημέρα λοιπόν κύριε Υπουργέ, κύριε πρέσβη, κύριε Φιούλε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, κυρία Συμπρόεδρε, κύριε... κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε περάσει πέντε χρόνια κοινών συνεδριάσεων και ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις έχουμε μπορέσει, στις δύσκολες εποχές έχουμε μπορέσει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας μέσα από τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Έχουμε περάσει μία περίοδο εκλογική, δημοκρατική, με ε, πολύ ξεκάθαρη έκφραση της θέλησης του λαού και θα ήθελα να απευθύνω το λόγο σε εσά, του ευρωβουλευτέ, που δυστυχώ δεν είσαστε πολύ άριθμοι εδώ παρόντε, δεν βλέπω πολλού ευρωβουλευτέ. Ε, ίσως αυτό να οφείλεται και στην εκλογική εκστρατεία ενώπιση των ευρωεκλογών, αλλά λυπούμε που δεν βλέπω μεγαλύτερη προσέλευση και παρουσία ευρωβουλευτών. Σας θα πρέπει στην προσεχή θητεία να γίνει μια προσπάθεια για περισσότερη ε, συμμετοχή των ευρωβουλευτών. Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω οι ευρωεκλογές να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και καλά αποτελέσματα συγκεκριμένα για τους συναδέλφους βουλευτές που είναι εδώ. Ε, οι κύριοι Τσαβούσογλου και Φιούλε θα καλύψουν ε, την ουσία των θεμάτων, γι' αυτό και εγώ τώρα θα σταματήσω και θα περάσω πάλι το λόγο στην συνάδελφο και συμπρόεδρο. Nous Ωραία. Αρχίζουμε λοιπόν ε, με τον ε, ε, Επίτροπο, τον Αρμόδιο για την Πολιτική Γειτονία και την Διεύρυνση. Δίνω το λόγο λοιπόν στον Στέφαν Φούλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας αγαπητοί συμπρόεδροι, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Καταρχάς, Η Ελέν Φλότρ είναι συμπρόεδρος αυτής της Επιτροπής τελευταία φορά. Θα ήθελα λοιπόν να σε επενέσω, ε, Ελέν, για την πολύ δραστήρια και επικοδομητική σου συμμετοχή στη δουλειά της Επιτροπής αυτής, όπως επίσης ε, και για την αμοιβαία ε, κατανόηση που προώθησες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Είναι η τελευταία μου ευκαιρία να σας μιλήσω. Δεν θα μπορούσε όμως να ήταν καλύτερη η χρονική στιγμή για την παρουσίαση των απόψεών μου για την κατάσταση των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κάνοντας πέντε παρατηρήσεις. Μέχρι το τέλος του 2013 ε, είδα ε, μια ανανεωμένη όθηση στις ε, σχέσεις μας, καταρχάς με το άνοιγμα του κεφαλαίου 22 για την περιφερειακή πολιτική. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας, διότι ανοίξαμε επιτέλους ένα νέο κεφάλαιο μετά από πάνω από τρία χρόνια και τώρα, επαφίεται στην Τουρκία να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία αυτή για να καθορίσει μία ε, περιφερειακή πολιτική που θα εμπνέεται από το ευρωπαϊκό μοντέλο. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι ε, τα μέσα προενταξιακής ενίσχυσης ε, έχουν υποστηρίξει την Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια. Δεύτερον, υπήρξαν ε, σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και της, και της δικαστικής εξουσίας. Τούρκοι οι πολίτες ε, βρίσκονται ενώπιον μιας πραγματικής ε, πιθανότητας ε, απελευθέρωσης των θεωρήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Για να μπορέσουμε να δρέψουμε τους καρπούς ε, αυτής της προσπάθειας, πρέπει η ε, συμφωνία να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν. Τα δικαιώματα των μεταναστών πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας. Είναι ένα σημαντικό ε, γνώμονας για να κρίνει κανείς την κατάσταση και την δυνατότητα απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Εγώ θα υποστηρίξω τις προσπάθειες αυτές. Τρίτον, Κατά τους τελευταίους μήνες ε, εξετάσαμε καλύτερα τις ε, εμπορικές μας σχέσεις, έγινε αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας ε, του Τελωνιακού Κώδικα, που είναι η ραχοκοκαλιά των σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας έδωσε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και όπως επίσης και τα ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Κα, καταρχάς μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το ε, δυναμικό ε, που παραμένει αναξιοποιητό ακόμα αν μπορέσουμε να υπερβούμε τις υπάρχουσες δυσκολίες. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τη συνεργασία μας για τα επόμενα έτη. Τέταρτη παρατήρηση. Είναι προφανές ε, ότι η επιτυχημένη συνεργασία ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας πρέπει να ε, βασιστεί και στην ενέργεια. Από κοινού τον Επίτροπο Έτιγκερ, εγώ υποστηρίζω στήριξα μια ενισχυμένη συνεργασία ε, βασισμένη σε ενεργειακό μείγμα με την Τουρκία, ε, όπως επίσης και την ανάπτυξη υποδομών, ε, την αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητά μας. Πέμπτη παρατήρηση, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουν τις προκλήσεις στην κοινή μας γειτονιά. Ε, οι προκλήσεις αυτές να αντιμετωπίζονται καλύτερα όταν συνεργαζόμαστε και επομένως και οι δύο πλευρές ε, εξακολουθούν να ενισχύουν τον στρατηγικό διάλογο και τη συνεργασία στην εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ε, στην ανανέωση ε, των, ε, συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Είχαμε λοιπόν με τον κύριο Παυτούγλου πάρα πολλέ συζητήσει τον Φεβρουάριο και είμαι πεπισμένο ότι θα υπάρξει ε, η δυνατότητα να ε, προωθήσουμε ακόμη περισσότερο τις συνομιλίες αυτές. Επίσης, έχουμε δει εξελίξεις και στον τομέα των διαδικασιών προσχώρησης, ε, οι οποίες δυστυχώς μας δημιουργούν ανησυχίες και απογοήτευση όσον αφορά το δικαστικό τομέα. Η νέα νομοθεσία ε, είχε ως αποτέλεσμα να περάσουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πολλές εξουσίες του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Τουρκίας, ε, κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα σε προηγούμενες μεταρρυθμίσεις που είχαν γίνει ε, με τη συνεργασία μας και δυστυχώς υπαναχωρεί σε σχέση με τις διεσμεύσεις που είχε λάβει η Τουρκία και στο Συμβούλιο, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και δημιουργεί ανησυχία σε σχέση με την ε, ε, αμεροληψία το, της δικαστικής εξουσίας και τη διάκριση των εξουσιών στην Τουρκία. Εκτός από τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις, ε, οι μεταθέσεις πολλών δικαστών, αστυνομικών αποτελούν ένα κίνδυνο για την σωστή ε, εκπόνηση έρευνας σε περιπτώσεις διαφοράς. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζονται και εξετάζονται οι ισχυρισμοί ε, ε, διαχείρισης και πρέπει να πω ότι με δυσαρεστεί η νέα νομοθεσία για το ίντερνετ δεν υπάρχει επαρκής προστασία, δεν υπάρχουν νομικά εχέγγυα ε, ε, διότι η πρόσφατη απαγόρευση των κοινωνικών μέσων ε, δείχνουν ότι οι ανησυχίες αυτές ε, δυστυχώς δικαιολογούνται. Υπάρχει σοβαρός περιορισμός της ελευθερίας έκφρασης, κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα σε σχέση με την αμεροληψία και την έκφραση όλων των απόψεων. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα γιατί κάθε περιορισμός θα έπρεπε να είναι αναλογικός, όπως προβλέπεται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Τουρκία μέσω της ε, εκθέσης προόδου μας ε, το φθινόπωρο. Πρέπει όμως να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Ειδικότερα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το τομέα του το, ε, κράτους δικαίου και των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να ενισχύσουμε το διάλογό μας σε όλους τους τομείς ε, πολιτικής και νομοθέτησης στον τομέα αυτό, που αποτελεί το επίκεντρο της διαδικασίας προσχώρησης. Πρέπει να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης πρέπει να συνεργαστούμε όσον αφορά την αξιολόγηση της ε, υφιστάμενης νομοθεσίας. Ως υποψήφια χώρα που έχει δεσμευθεί στο να προωθήσει τη διαδικασία προσχώρησή της, η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει, να έχει πλήρη γνώση των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βέλτιστων πρακτικών της. Τι σημαίνει αυτό τώρα ε, σε πιο συγκεκριμένα. Πρέπει να έχουμε ένα θετικό ε, πρόγραμμα ε, συγκεκριμένα στον τομέα της ομάδας εργασίας για το κεφάλαιο 23. Επίσης, τακτική πολιτική παρακολούθηση σε τεχνικό επίπεδο θα πρέπει να συμπληρώνει τον διάλογό μας κάτι το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το δυναμικό των ε, φορέων, των ε, υποεπιτροπών, ε, το, της Επιτροπής Σύνδεσης και του Συμβουλίου Σύνδεσης που αποτελούν πυλώνες της συνεργασίας μας. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία της επερχόμενης αξιολόγησης ομοτήμων για να ενισχύσουμε τη συνεργασία, γιατί έχουμε αποφασίσει ήδη με τις τουρκικέ αρχές να έχουμε μία αξιολόγηση ομοτήμων για την ελευθερία της έκφρασης. Αυτή η αξιολόγηση θα μπορούσε να εξετάσει λεπτομερώς τα ζητήματα όπως η εφαρμογή της νέα νομοθεσία που αφορά το διαδίκτυο. Στο ε, τρέχον πλαίσιο η συνεργασία των τουρκικών αρχών ε, στο πλαίσιο του εγχειρήματο αυτού είναι εξαιρετική σημασία. Το ίδιο ισχύει και για, τις, ε, για την αξιολόγηση ομοτήμων ε, για το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων, όπως επίσης και για το ποινικό και δικαστικό σύστημα. Θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την, την αμεροληψία, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία. Είναι, αποτελ, απο, είναι βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο ε, μια στρατηγικής σχέσης. Δημιουργούνται ε, παρεξηγήσεις, δημιουργούνται διαφωνίες και μια καλύτερη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές ε, θα μας επιτρέψουν να φέρουμε την Τουρκία πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μεταρρυθμίσεις να μην έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει, πάντοτε ήταν υπέρμαχος της ε, προώθησης ε, των, ε, της διαδικασίας προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμως να είμαστε να συνεργαζόμαστε και να είμαστε ειλικρινείς. Τα, οι τελευταίοι μήνες και οι τελευταίες εξελίξεις έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες σε σχέση με τις προδιαγραφές και τη στάση της Τουρκίας και ελπίζουμε ότι κατά τους επόμενους τρεις μήνες θα διαψευστώ ε, ότι η Τουρκία θα δεσμευτεί ενέου, ε, εκ νέου ε, για την, τις μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν τη χώρα σας πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επικοδομητική συνεργασία θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό μας, των σχέσεών μας, πλήρως και ε, να είστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να σας βοηθήσει στην προσπάθεια σας αυτή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πάντα μετρημένα μιλάτε. Με τοποθετήσεις προσεκτικές που δείχνουν ότι είστε πραγματικό φίλο τη Τουρκία, Κύριε Πρέσβη, εκ μέρου τη ε, ελληνική προεδρία, ο κύριο Σωτηρόπουλος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φλότρ, αγαπητοί συμπρόεδροι, ε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, ε, αγαπητέ Σελίμ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Προεδρίας θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή που μου δίνει τη δυνατότητα να σας πω μερικά λόγια για το ύψιστη σημασία σημασίας θέμα ε, των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωση και Τουρκίας. Η συνεδρίασή μας ε, ε, λαμβάνει χώρα σε μια σημαντική χρονική στιγμή. Ελλάδα είναι και ήταν πάντοτε υπέρμαχος ε, της ε, ε, διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν γίνει αλλαγές από την προηγούμενη ελληνική προεδρία και την Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης του 2013 οι εξελίξεις δείχνουν ε, την, ε, το σταθεροποιητικό αποτέλεσμα της διαδικασίας της διεύρυνσης. Θα ήθελα τώρα να τονίσω τη σημασία που δίνει το Συμβούλιο στις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η Τουρκία είναι και υποψήφια χώρα και βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μας ενεργεί, ενεργεί και ε, συνεχή συνεργασία ε, με πλήρη σεβασμό όλων των ε, προϋποθέσεων της διαδικασίας προσχώρησης θα δώσει τη δυνατότητα στην Τουρκία να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της. Ε, οπότε επικροτούμε το άνοιγμα του κεφαλαίου 23 για την περιφερειακή πολιτική και το συντονισμό των διαδροτικών μέσων ε, που ανανεώνει ε, τις, τις σχέσεις Ευρω... Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θα ήθελα να πω ότι εμείς παραμένουμε δεσμευμένοι να βοηθήσουμε την Τουρκία στην προσπάθειά της από τη στιγμή βέβαια που οι απαιτήσει πληρούνται. Είναι σημαντικό η Τουρκία να χρησιμοποιήσει όλες τις ευκαιρίες για περαιτέρω πρόοδο στις διαδικασίες προσχώρησης. Αυτό βέβαια χρειάζεται πολιτική βούληση και στένος, αλλά είναι προς όφελος όλων. Ο ρυθμός των διαπραγματεύσεων μπορεί να επισπευθεί αν η Τουρκία προχωρήσει ε, στην πλήρωση των ε, των ορόσημων ε, ώστε να πληρεί τις απαιτήσεις του διαπραγματευτικού πλαισίου. Οπότε καλούμε την Τουρκία να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να ανοίξουν ε, το, για να ανοίξει το κεφάλαιο 5, δημόσιες συμβάσεις, 8 ε, ε, ανταγωνισμός και 19 κοινωνική πολιτική και ασφάλεια. Επίσης πρέπει να εφαρμοστεί το επιπλέον πρωτόκολλο για την ε, συμφωνία σύνδεσης, όπως επίσης ε, και την ε, ομαλοποίηση των σχέσεων της Τουρκίας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Κάτι το οποίο θα ενισχύσει την την πρόοδο των διαδικασιών διαπραγμάτευσης. Ε, η Τουρκία πρέπει να προχωρήσει ειδικότερα στον τομέα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και το Συμβούλιο εξακολουθεί να ενθαρρύνει την Τουρκία να ε, κάνει μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν ε, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και των μειονοτήτων. Η εφαρμογή βάσει ευρωπαϊκών προτύπων είναι σημαντική. Επίσης το Συμβούλιο λαμβάνει γνώση και βλέπει θετικά την ανάπτυξη της ενεργού κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία που πρέπει να υποστηριχθεί και να θεωρηθεί ένας ε, ένας ε, σημαντικός και ε, θεμητός εταίρος. Επίσης, χαιρόμαστε όλος ιδιαίτερος με την ύπαρξη του διαμεσολαβητή και άλλων θεσμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα χρειαστούν όμως ιδιαίτερες προσπάθειες σε σχέση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων και των, ε, της ελευθερίας ε, στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε, του συναστρίζεστε, ε, της έκφρασης, της ελευθερίας θρησκείας, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η χρήση επίσης υπερβολικής βίας είναι κάτι που πρέπει να ε, ερευνηθεί. Οι περιορισμοί ε, στα ε, μέσα τα κοινωνικά, όπως προσφάτως του Twitter και του YouTube είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει ε, όπως επίσης και το γεγονός ε, ότι διώκονται ε, προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι. Θα ήθελα επίσης να σας πω ε, ότι στις 20 Ιανουαρίου ε, επισκέφθηκαμε τον Πρωθυπουργό Ερντογάν, ε, ο οποίος συναντήθηκε με τον Φαντρόμπα, τον, Παρόσο, τον κύριο Παρόσο και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Σούλτς. Υπήρξαν ανησυχίες σε σχέση με τη διάκριση των εξουσιών, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της δικαστικής εξουσίας, όπως επίσης και μιας πραγματικής δικαστικής έρευνας και σωστής έρευνα σε σχέση με ε, ισχυριζόμενη κακομεταχείριση και επαγγελματική αμέλεια ε, πρέπει να υπάρξει νέα νομοθεσία ειδικότερα σε σχέση με το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και ενισχύει τον έλεγχο της κυβέρνησης στη δικαστική εξουσία. Ε, πρέπει να ε, η Τουρκία να δείξει ότι δεν υπαναχωρεί, ότι παραμένει δεσμευμένη ε, στην πλήρωση των όρων της διαδικασίας προσχώρησης και πρέπει να επιτρέψει τη δικαστική εξουσία να λειτουργήσει με αμερόληπτο και ανεξάρτητο τρόπο. Πρέπει να δείξει ότι παραμένει δεσμευμένη στο σεβασμό των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Επίσης οι κοινωνικές ε, συνθήκες ε, για τις δίκες ε, είναι κάτι το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην Τουρκία να σεβαστεί τις απαιτήσει των ίδιων των πολιτών της. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί της, την, συμφωνία της, την, την υπογραφή της Συμφωνίας Επανεισδοχής ο διάλογος ε, για την απελευθέρωση των θεωρήσεων θα βασιστεί στις επιδόσεις της Τουρκίας, ε, όπως επίσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής των απαιτήσεων που υπάρχουν στον οδικό χάρτη, ε, όπως αυτός εγκρίθηκε στο, από το Συμβούλιο. Όσον αφορά τώρα την ε, παράνομη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η ύπαρξη των διμερών συμφωνιών επαντησδοχής ε, είναι κάτι το οποίο παραμένει προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό η νομοθεσία για τη διεθνή προστασία των αλλοδαπών είναι μια σημαντική πρόοδο στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Στον τομέα τώρα της εξωτερικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία έχουν θετική συνεργασία. Υπάρχουν πολλές ε, συνεδριάσεις ε, όσον αφορά τη Συρία, το Ιράν, την Ουκρανία, την, Αίγυ... την Αίγυπτο, τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, μεταξύ άλλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει ε, τις αποστολές στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ ε, ώστε να βοηθήσει ε, τη συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ώστε να υπάρξει ευθυγράμμιση με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση με τα προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επιμένει η Τουρκία να προβεί σε ειρηνική επίλυση διαφορών, οπότε κάνει έκκληση στην Τουρκία να αποφύγει απειλέ ή ε, δράσει εναντίον κρατών μελών ή ε, κοινωνική ρήξη που θα μπορούσε να διαταράξει τις ε, καλέ καλές γειτονικές σχέσεις και την ειρηνική επίλυση διαφορών πρέπει να υπάρχει σεβασμός όλων των προϋποθέσεων, δηλαδή διμερείς συμφωνίες και σεβασμός του κοινοτικού κεκτημένου. Ε, όπως επίσης το σεβασμό των ε, κυρίαρχων δικαιωμάτων ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να γίνουν σεβαστά από την Τουρκία. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να οδηγήσουν τις συνθήκες για την επίλυση την ειρηνική του κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στους οποίους βασίζεται η συνεργασία μας με την Τουρκία για αυτό το θέμα. Ε, η δέσμευση της Τουρκίας ε, θα ε, είναι κρίσιμη και θα μπορούσε να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό των διαπραγματεύσεών μας με την Τουρκία. Ελπίζω ότι κατά τους επερχόμενους μήνες θα υπάρξουν καλύτερες εξελίξεις στη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, επικεφαλής διαπραγματευτά εκ μέρους της Τουρκίας. Κύριε Τσεγούσογλου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Συμπρόεδρε. Αγαπητέ φίλε, κύριε Φίλε, αξιότιμη πρέσβης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από την ευρωπαϊκή πλευρά αλλά και από την τουρκική πλευρά Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή και για την ευκαιρία να συζητήσουμε. Για μένα είναι η πρώτη, αλλά και η τελευταία συνεδρίαση αυτής της θητείας για την Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή όπου συμμετέχω. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την υποστήριξη την οποία έχει προσφέρει στη διαδικασία για την ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, συμπρόεδρο κυρία Φλότρο για την προσωπική υποστήριξη που έχει προσφέρει στην υπόθεση αυτή, αλλά και την κυρία Όμεν Ρόιτεν, την εισηγήτρια τη εκθέσεω για, την, ε, για την πρόοδο τη Τουρκία. Θέλω να σα ευχαριστήσω λοιπόν και τι δύο ιδιαίτερω. Εμεί είτε στι σχέσει ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, την, και το Συμβούλιο είτε εδώ έχουμε ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή πάντοτε οποιασδήποτε επικρίσεις έχουν διατυπωθεί και τις ε, ακούμε με πολύ μεγάλο σεβασμό διότι πιστεύουμε ότι έχουμε έναν φυσικό σύμμαχο στο πρόσωπό σας, στο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη διαδικασία και ότι ο κοινός στόχος είναι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι μας βοηθάτε να προχωρήσουμε στη διαδικασία αυτή με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο ε, χωρίς εμπόδια. Βεβαίως υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν, υπήρξαν πολιτικά προσκόμματα, ε, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σήμερα σε αυτά, αλλά υπάρχουν στο παρελθόν μα είτε ήταν η Κύπρο, είτε ήταν άλλοι λόγοι. Κάποια κράτη βρήκαν ε, μέσω τη επιτροπή τη δυνατότητα να παρεμποδίσουν την ε, πρόοδο των σχέσεών μας. Δεν πρέπει να μα επηρεάζουν όμω αυτά. Ο κύριο Φίλε το είπε, το Συμβούλιο Συνδέσεως και οι πολιτικές πλατφόρμες, οι επιτροπές, οι υποεπιτροπές που συστήνονται, συζητούν ε, είτε τη δυνατότητα για άνοιγμα των κεφαλαίων, είτε και αν δεν μπορούν επίσημα να ανοίξουν τα κριτήρια γιατί δεν προβλέπονται, τα κεφάλαια γιατί δεν προβλέπονται τα κριτήρια, δεν επαρκούν τα κριτήρια την ανεπίσημη συζήτησή τους. Ε, εμείς έχουμε μπορέσει λοιπόν χάρη σε όλα αυτά να προχωρήσουμε σε μια πορεία προόδου η οποία αποτελεί προσαρμογή στα κριτήρια της ένταξη και τα κεφάλαια, χωρίς όμως απαραίτητα να σημαίνει αυτό ότι έχουμε περάσει τη διαδικασία του ανοίγματο. Δηλαδή συνεχίζουμε εμείς μα εσωτερικά, ανεξαρτήτως του τι υπαγορεύουν τα κεφάλαια, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι καλό για τη χώρα. Έχουμε λοιπόν ένα, μια θετική εξέλιξη από το 2013 με το άνοιγμα του 22ου κεφαλαίου για την περιφερειακή πολιτική. Έχουμε μια θετική εκτίμηση από την έκριση της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργό μας ε, άλλωστε ανακοίνωσε και το πακέτο του εκδημοκρατισμού. Το 2013 λοιπόν ως έτος προς το τέλος βλέπει την υπογραφή της Συμφωνίας για την Επανεισδοχή και την, ε, και την εκκίνηση της ε, απαλλαγής από την υποχρέωση των διαβατηρίων για τους Τούρκους Επικού. Έχουμε λοιπόν μια θετική ε, τάση η οποία επιβεβαιώνεται πιστεύω το 2014. Στις αρχές του χρόνου ο Πρωθυπουργό μας το δήλωσε. Το 2014 θα είναι έτος καμπής για τι σχέσει τη Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζουμε και εντείνουμε τι διπλωματικέ μα επαφέ είτε στι Βρυξέλλε, είτε στο Βερολίνο, είτε στην Ιταλία, τη Δανία, την Ουγγαρία. Μια σειρά λοιπόν χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδέχθηκαν είτε τον ε, Πρωθυπουργό μας, είτε ε, τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και έχουμε ως βλέπετε μια εντατικοποίηση των σχέσεων. Ο δε πρόεδρος της Γαλλίας ήρθε και επισκέφθηκε ως πρώτος ύστερα από 22 χρόνια Γάλλος Πρωθυπουργός την Άγκυρα σε μια συμβολική κίνηση. Από όλα αυτά προκύψει ένα πολύ σαφές αποτέλεσμα. Ότι τώρα πρέπει να πατήσουμε τον γκάζι στις διαπραγματεύσεις, να επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις και να τις αντιδικοποιήσουμε. Ιδιαίτερα τα κεφάλαια 22 και 23 πρέπει να ανοίξουν το ταχύτερον δυνατό. Είναι κάτι το οποίο εμείς υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα. Είναι τα κεφάλαια που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι τα κεφάλαια που έχουν να κάνουν με την, ε, το 23 και 24, συγγνώμη, με τη δικαιοσύνη της ελευθερίας και την ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, πιστεύουμε ότι πρέπει να ανοίξουν το χειρότερο δυνατό. Ε, έχουμε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την κυρία Μέρκελ συγκεκριμένα και από άλλους ε, πολύ σαφείς τοποθετήσεις. Δυστυχώς όμως η, η ελληνοκυπριακή διοίκηση για πολιτικούς λόγους παρεμποδίζει το άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών, λέει ο μιλητής, και θα πρέπει να δούμε ποιον πρέπει να πείσουμε. Τώρα οι φίλοι και γη των Ελλάς είναι εκείνοι που θα πρέπει να πιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που θα πρέπει να πιστεί. Οι χώρε μέλη χωριστά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με πρώτε πρώτε τη Γαλλία και η Γερμανία. Προ αυτέ πρέπει να στραφούμε. Για να ανοίξουν λοιπόν τα κεφάλαια αυτά, εμεί οπωσδήποτε θέλουμε να ανοίξουν και θέλουμε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει σε αυτά τα θέματα δε, ο δε πρόεδρο τη Ρουμανίας, Μπασέσκου, σε μια επίσκεψη στην Τουρκία μα είπε ξεκάθαρα ότι, πρέπει, ότι θέλουν να ανοίξουν τα κεφάλαια, ότι του ενδιαφέρει προσωπικά διότι είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει, παρότι έχουν καταστεί εδώ και τόσα χρόνια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διαπραγματεύσει τα κεφάλαια αυτά. Του ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ, βλέπουν πόσο σημαντικό είναι. Προϋποθέση ωστόσο ε, για κράτη που αρχίζουν το τελευταίο διάστημα τη διαπραγματεύση είναι πρώτα να ανοίξουν και να κλείσουν τα κεφάλαια αυτά. Έχει αλλάξει δηλαδή η σειρά και η προτεραιότητα. Εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε ω Τουρκία, το καθήκον μα και πιστεύουμε ότι το 2014 θα είναι ένα έτο μεταρρυθμίσεων. Πιστεύουμε ότι το 2014 ξεκίνησε με διαπραγματεύσει και θα συνεχίσει διαπραγματεύσει. Γιατί ήταν η νομοθεσία για το ίντερνετ. Είτε ήταν το ζήτημα της, ε, των αλλαγών στην νομοθεσία τη σχετική με τους δικαστές και εισαγγελείς και οι σχετικές αντιπαραθέσεις. Είτε ήταν το θέμα του Twitter και των, ε, ε, κοινωνικών δικτύων. Ακούσαμε τα σχόλια και τις επικρίσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θέλουμε να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα δράσης με τη σειρά που αναφέρεται. Η, η σειρά προβλέπει και το θέμα των δικαστών και εισαγγελέων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προβλέπεται από τα μέτρα που εμείς προτείνουμε να διευρυνθούν και να ε, ενισχυθούν. Στο πακέτο μέτρων για τη δικαιοσύνη έχουμε μπορέσει και μάλιστα μέχρι την τελευταία στιγμή πριν χρειαστεί να κλείσει η Βουλή εν ώψη των τοπικών και περιφερειακών εκλογών, δηλαδή μέχρι ε, ώρα εκ της πρωινής και 6 λεπτών πριν να κλείσει η Βουλή την τελευταία στιγμή, δούλευε το Κοινοβούλιο μας για να εγκρίνει την νομοθεσία, για να εγκρίνει αυτό το δικαστικό πακέτο το οποίο έχει ε, φέρει σημαντικές μεταρρυθμίσεις ως προς το θέμα της ε, αντιμετώπισης των τρομοκρατικών πράξεων, ω προς το ζήτημα της του δικονομικού ποινικού δικαίου και πολλά άλλα. Έχει εξασφαλίσει πολύ καλύτερη ε, μεταχείριση δικαστική των κατηγορουμένων έχει μειώσει στα 5 από 10 χρόνια την περίοδο της προσωρινής κράτησης για συγκεκριμένα δικήματα και ε, θέλω να επισημάνω εν προκειμένου ότι παρότι εμεί είχαμε κοινοποιήσει αυτέ τι μεταρρυθμίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπουμε με λύπη ότι δεν περιλήφθησαν στην έκθεση προοδού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι κάτι όμω το οποίο με χαρά διαπιστώνω πώ θα συζητήσουμε και σήμερα αύριο σε αυτή μα την διημερή συνεδρίαση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε όλα τα θέματα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Η ενέργεια, παραδείγματι, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με την άτυπη σύνοδο των Υπουργών των Εξωτερικών στην Αθήνα, στην οποία είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω, δόθηκε η έμφαση στην ενέργεια και την εξάρτηση από τη Ρωσία πολλών κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στο πώ μπορούμε να απεξαρτηθούμε από αυτή την εξάρτηση από την προμήθεια ενέργεια τη Ρωσία. Είναι κάτι που μας απασχολεί και εμάς ιδιαιτέρως. Για το 15ο όμως αυτό κεφάλαιο της ενέργειας, το ότι δεν ανοίγει το κεφάλαιο αυτό για την Τουρκία, δυστυχώς ε, λυπούμαστε πάρα πολύ, πρέπει να εκφράσουμε τη λύπη μας. Ο κύριος Φίλε έχει κάνει τις προσπαθειές του, αλλά δεν έχει επιτύχει να ξεκινήσει το άνοιγμα. Θέλουμε επίσης να συμμετέχουμε είτε πρόκειται για θέματα εξωτερικής πολιτικής είτε πρόκειται για θέματα της εγγύης γειτονίας στις συνεδριάσεις του, Υπουργείου, του Συμβουλίου των Εξωτερικών στις άτυπες ιδιαίτερως θέλουμε να είμαστε παρόντες δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν μας επιτρέπεται η συμμετοχή όταν έχουμε να κάνουμε την εξωτερική πολιτική όταν έχουμε να κάνουμε με την Ουκρανία και τη Ρωσία και τις σχέσεις με τις χώρες αυτές όταν εξετάζονται αυτά τα σοβαρά θέματα Βλέπουμε άλλωστε τις ανεπάρκειες που πληρώνει τώρα η Ουκρανία αυτής της πολιτικής. Δεν έχει κανένα δικαίωμα, δεν έχει καμία, κανένα νόμιμο έρισμα η Ρωσία στα όσα πράττει. Εμείς όμως θέλουμε να είμαστε σε θέση μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσουμε πού είναι τα δικά μας φάλματα, πού ήταν οι δικές μας οι ελλείψεις και τα υστερήσεις και πώς θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερα ε, βοηθήσει την Ουκρανία γιατί δεν έχουμε πολυτέλεια να ε, αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ε, γεγονότα και στο μέλλον ή να διονυστεί αυτό το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε και να παραδεχθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι είδους ευθύνες έχουμε ή συνυπευθυνότητα έχουμε για το θέμα αυτό. Ε, ένα θέμα που έχουμε ας πούμε με την Αρμενία, την υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας που έχει να κάνει με τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Πόσο έχουμε βοηθήσει, πόσο έχουμε παρεμποδιστεί και από τη Ρωσία που σε τελευταία ανάλυση και με τη Μολδαβία βλέπουμε τη στάση έχει τηρήσει και με το θέμα της Κύπρου που θέλω να επισημάνω ιδιαίτερος, διότι ευτυχώς είπε ο κύριος Φίλε ξεκινάνε νέες συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού. Η Ελλάδα ξέρουμε ότι και εκείνη συμφωνεί ότι πρέπει να προχωρήσει το θέμα αυτό. Ε, ας μην χάσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό να λυθεί το θέμα αυτό με μία λύση που θα είναι κερδισμένες και οι δύο πλευρές. Νομίζω ότι το θέμα αυτό πρέπει να επισημάνω, το Κυπριακό, παρότι είχαμε εσωτερικέ δημοκρατικέ και τοπικέ εκλογέ στην Τουρκία, δεν κατέστη αντικείμενο λαϊκισμού και ε, εκμετάλλευση για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και αυτό πρέπει να εκτιμηθεί και να μπει στα θετικά τη Τουρκία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τι προσπάθειέ μα και θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του Ανώτατου Συμβουλίου Εισαγγελέων και Δικαστών που ανέφερε ο κύριο Φιούλε και τη σχετική απόφαση. Εμεί ω Τουρκία εγγυόμεθα την εσωτερική και εξωτερική ανεξαρτησία και ασφάλεια των δικαστών και εισαγγελέων στο λειτουργήμά του. Υπάρχουν αποφάσεις των και, των εισαγγελέων και δικαστών, συγγνώμη, οι οποίες δεν ε, είναι καθόλου ευχάριστη στην κυβέρνηση, παρόλα αυτά όμω δεν παρεμβαίνει και αυτό αποτελεί νομίζω κατάφορη απόδειξη τη ανεξαρτησία του δικαστικού και εισαγγελικού σώματο. Πάντω για την ε, πορεία αυτή τη μεταρρύθμιση με τη σχετική νομοθεσία πρέπει να επισημάνω ότι δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έφερε το θέμα αυτό στην επικαιρότητα τη συζητήσεώ του. Εμεί ενημερώσαμε τον κύριο Φιούλε ε, βήμα το βήμα για την κάθε πορεία, για το κάθε άρθρο όπω προχωρούσαν οι μεταρρυθμίσει. Κάναμε προτάσεις, ακούσαμε συστάσεις, ακολουθήσαμε από τις 8 τις 5, από τις 8 ε, τις άλλες 2 τις δεχθήκαμε εν μέρη και προσαρμόσαμε αναλόγως την νομοθεσία μας και άρα εισήχθησαν οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει λοιπόν συνεργασία, αυτό ήθελα να πω και εν τέλει θα θέλαμε και εμείς να επαναλάβουμε μία σύσταση που έχουμε ήδη διατυπώσει, ότι δηλαδή θα πρέπει να επανεξεταστεί και να αντιπαραβληθεί αυτή η νομοθεσία της Τουρκίας και στο πρώτο της καρύφωμα αλλά και στην τελική της μορφή με την αντίστοιχη νομοθεσία που ισχύει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί νομίζω ότι η δική μας νομοθεσία εάν αντιπαραβληθεί θα, θα αποδειχθεί πολύ πιο φιλελεύθερη και πιο ε, δημοκρατική. έχουμε πει ξεκάθαρα στον κύριο Φιούλε. Είναι μια πρόταση την οποία επαναλαμβάνουμε και πάλι. Οι υπουργοί μας, πρωθυπουργοί, βασιλείς, μου απαντήσατε, έχουν θέματα εσωτερικής πολιτικής, δεν μπορούν να γίνουν όργανα για την ε, ε, σύγκριση της νομοθεσίας Τουρκίας, δεν έχουμε τη σχετική αρμοδιότητα για να επαληθεύσουμε τα ε, την εσωτερική νομοθεσία των κρατών μελών, μου λέτε κύριε Φιούλε. Όμως έχετε αντίστοιχα την δυνατότητα να επαληθεύεται και μάλιστα με πολύ μεγάλη δυσπιστία την ε, εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας. Αυτό είναι το δυστύχημα. Λυπούμε πάρα πολύ. Ήμασταν υποχρεωμένοι να διατυπώσουμε αυτή μας τη δυσαρέσκεια ξεκάθαρα στους φίλους μας. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις η Τουρκία. Έχουμε μία σειρά από που θεσπίσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για, την, για το δικαίωμα ατομικής προσφυγής στο συνταγματικό δικαστήριο, που σημαίνει και μείωση του φόρτου εργασίας και του συνταγματικού δικαστηρίου, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε θέσπιση του διαμεσολαβητή, του, του ε, εκπροσώπου του πολίτη, του Ombudsman δηλαδή, ε, έχουμε μια σειρά από νομοθεσίες από νομοθετήματα, από νομοθετήματα τα οποία έχουν προχωρήσει όπως είπαμε, ιδιαίτερα τα θέματα της παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ε, περιβολικά μακρά προσωρινή κράτηση και πολλά άλλα, είναι ζητήματα τα οποία έχουν και αντιμετωπιστεί νομοθετικά, αλλά και οδηγήσει σε αποζημιώσει περίπτωση παραβιάσεως των, δικαιωμάτων προς τους συγκεκριμένους παθόντες. Για το ίντερνετ και τα κοινωνικά θέματα θα ήθελα να σας πω τα εξή. Εμείς ως ε, Υπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων αλλά και παλιότερο όταν είχα την Προεδρία του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης δεν είναι δυνατόν εγώ προσωπικός να παραγνωρίζω τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα ωστόσο να πω ότι το κύριο θέμα και το βασικό θέμα για μένα είναι το εξή. Ότι η ελευθερία τη έκφραση, η ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση, η ελευθεροτυπία δεν μπορεί στο όνομα της διαφύλαξης κάποιων ανθρωπίνων δικαιωμάτων να παραβιάζει την ε, ιερή ιδιωτική ζωή, τον ιδιωτικό βίο. Δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα δηλαδή. Εμείς έχουμε κάνει με τις ε, μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και την, ε, έχουμε εξασφαλίσει και την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του ιδιωτικού βίου. Αυτά είναι θεσπισμένα, θεσμοθετημένα στην νομοθεσία μας. Έχουμε επίσης και από τη συμφωνία, Διεθνή Συμφωνία για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα εγγυηθεί το απόρριτο του ιδιωτικού βίου και το ε, απρόσβλητο του ιδιωτικού βίου είναι κάτι το οποίο, ε, στο οποίο δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και καταλαβαίνετε ότι όταν γίνονται παράνομες παρακολουθήσεις ε, μυστικών συνεδριάσεων στις οποίες συμμετέχει ο Υπουργός των Εξωτερικών δεν είναι δυνατόν να τις παραγνωρίζουμε και να μην λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Ήδη το 1970 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης είχε κάνει συστάσεις και αργότερα κάποιες άλλες, οι οποίες στείλουν προς την ίδια κατεύθυνση. Μέχρι και την τελευταία του 2012, η οποία πάλι μιλάει για την προστασία του ιδιωτικού βίου των ιδιωτών και τη δυνατότητα προστασίας από παραβιάσεις αυτού του ιδιωτικού χώρου. Αυτό λοιπόν είναι η αναζήτησή μας, αυτή η ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας του λόγου και του απόρριτου του ιδιωτικού βίου, η κρίση του τι είδου μέτρα επιβάλλονται, της ποιότητας των μέτρων που επιβάλλονται, πάντα θα έχει να κάνει με την βαρύτητα και την αναλογικότητα σε σχέση με την παραβίαση. Εμείς είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε πρόκειται για την ε, Επιτροπή της Βενετίας. Με πολύ μεγάλη προσοχή ακούμε τις συστάσεις σας, τις παρακολουθούμε και αναλόγως κάνουμε την προσαρμογή της νομοθεσίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνουμε ότι Πραγματικά ε, ε, σας ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, η δουλειά του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μας το δείξατε και στην ομιλία σας, το γνωρίζαμε και από πριν. Να δώσω το λόγο καταρχάς στην κυρία Όμεν Ρόιτεν. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, ακύρωσα μόλις μία συνεδρίαση ε, του Ιδρύματος Φρίντριχ ε, Έμπερτ, γιατί νόμιζα ότι η σημερινή συνεδρίαση ε, είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι σημαντικό για μένα να είμαι εδώ για να εκφράσω την άποψή μου. Ειδικότερα είναι και η τελευταία συνεδρίασή μου πριν από τις ε, εκλογές, γιατί μετά τις εκλογές ε, ο Ήρο Λέινας θα είναι υποψήφιος για τη δική μου θέση και γνωρίζει την Τουρκία πολύ καλά και μιλάει και τουρκικά πολύ καλά. Στην Επιτροπή ΑΦΕΤ αλλά και στην ε, ε, Ολομέλεια υπήρχε μια πολύ αρνητική στάση, μια πολύ αρνητική διάθεση. Από το 2007 είμαι υπεύθυνη για την πρόοδο της ε, Τουρκίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μου Ε, προσπάθεια ήταν ένας ε, απόλυτα ανοιχτό διάλογος με την Τουρκία. Βάσει αυτού του διαλόγου εκπονήσαμε τις εκθέσεις μας και προσπαθήσαμε τουλάχιστον να πείσουμε ο ένας τον άλλον. Πριν από το 2007 ε, έβλεπα συχνά στις ε, συνεδριάσεις μας ε, και στις πολιτικές μας ομάδες ότι υπήρχαν προκαταλήψεις που επηρέαζαν τις πολιτικές απόψεις και από το 2007 και μετά προσπάθησα να έχουμε αυτόν τον ανοιχτό πολιτικό διάλεκτο, ε, διάλογο. Επίσης αυτό προσπάθησα να κάνω είναι να πείσω τους ε, Ευρωπαίους πολίτες ε, ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι είναι σημαντική χώρα. Επίσης προσπάθησα να τους πείσω ότι ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους πολίτες της Τουρκίας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και για τους ε, Τούρκους πολίτες αλλά και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί αν η Τουρκία αποτελέσει μια ευημερούσα σύγχρονη χώρα είναι καταρχάς σημαντικό και για τους ε, ε, Τούρκους πολίτες αλλά και για τους δικούς μας πολίτες. Αυτό που επίσης έκανα από το 2007 και μετά, θα ήθελα ειδικότερα να αναφερθώ στο έτος 2010 σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις ε, του δικαστικού τομέα, τις επικροτήσαμε, τις ενισχύσαμε, τις μεταρρυθμίσεις αυτές και αν δω τώρα πώς έχουν τα πράγματα, πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι απογοητευμένη. Είμαι πραγματικά απογοητευμένη. Όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί συνάδελφοί μου που δεν μπορούσαν ε, να ε, προβλέψουν αυτό που συνέβη. Όλοι υπερασπιστήκαμε τις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι αντί να συνεχιστούν να εξελιχθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, περιορίζονται περαιτέρω οι εξουσίες του δικαστικού τομέα απαγόρευση του Twitter, για παράδειγμα, απαγόρευση του YouTube. Είδαμε ότι το συνταγματικό δικαστήριο είπε ότι η απαγόρευση είναι απαράδεκτη. Και μετά είδα, διάβασα ότι θα έπρεπε να μειώσουμε τις εξουσίες του, του συνταγματικού δικαστηρίου. Μα δεν είναι δυνατόν να δουλεύει έτσι ε, μια δικαστική εξουσία. Σε ένα κράτος δικαίου υπάρχει διάκριση των εξουσιών, αυτό είναι το ένα πράγμα. Από την άλλη όμως, πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το κράτος δικαίου και αν λειτουργεί. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη διάρθρωση του κράτους δικαίου για πολιτικούς λόγους. Το κράτος δικαίου είναι αυτό που είναι και αν μία πολιτική πλευρά διαφωνεί, αυτό δεν θα έπρεπε να καταστρέφει το κράτος δικαίου. Εκεί είναι το πρόβλημα και νομίζω ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες, ο ρόλος ε, μιας αμερόληπτης ανεξάρτητης δικαστικής ε, ε, εξουσίας. Εμείς προτείναμε να ανοίξουν τα κεφάλαια, αλλά δεν χρειάζεται να ανοίξουν τα κεφάλαια, γιατί αν δει κανείς τα κριτήρια της Κοπενχάγης, ούτως ή άλλως ξέρετε ποια είναι τα ορόσημα και τι πρέπει να κάνετε. Οπότε το ίδιο ισχύει για την ενέργεια. Εγώ δεν διαφωνώ να τα ανοίξουμε τα κεφάλαια, αλλά δεν χρειάζεται, μπορείτε να προχωρήσετε με τις ε, μεταρρυθμίσεις, αν το θέλετε. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Και ο Επίτροπος, ο Στέφαν Φιούλε, μας είπε ότι είναι απογοητευμένος. αν δεν ανανεώσετε τη δέσμευσή σας, αν δεν υπάρχει και πάλι μία αμοιβαία προσήλωση ε, στους στόχους, στους επόμενους μήνες, γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να πέσουν λίγο οι τόνοι, να μειωθεί η έντοση στη χώρα σας, γιατί όλα αυτά τα πράγματα ε, θα γίνουν πολύ χειρότερα λόγω της ε, προεκλογικής περίοδου εν ώψη των εκλογών. Γι' αυτό ακριβώς εγώ ακύρωσα τη συνάντησή μου σήμερα για να είμαι εδώ. Ελπίζω, αυτό θέλω να σας πω, ότι με το επόμενο κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όπως κάναμε και από το 2007 και μετά. Το ελπίζω πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εκφράσατε πολύ καλά την άποψη των ε, συναδέλφων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ελπίζω ότι και στο επόμενο Κοινοβούλιο θα είναι εξίσου σημαντικός ο αριθμός των συναδέλφων που δεν έχουν κανέναν ενδιασμό σε σχέση με την ενίσχυση της ε, διαδικασίας προσχώρησης της Τουρκίας. Πραγματικά είπατε απογοητευμένοι, να μην πω ανήσυχοι για την κατάσταση. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, γιατί αυτό που φαίνεται να γίνεται υπό την πίεση των εξελίσεων και των γεγονότων, ε, ο δρόμος που ακολουθείται αυτή τη στιγμή μας φαίνεται επικίνδυνος. Ο κύριος Σαΐν και μετά ο κύριος ε, Νταφ. Ε. Ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω και να χαιρετήσω τον κύριο Φίλιο, τον κύριο Τσόουσουγλου, τον, ε, τους ε, δύο πρέσβες, την εισηγήτρια, κυρία Ομεν Ρόιτεν για τις αντιφέρουσες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις. Μιλήσατε για απογοητεύσεις στη σχέση με την Τουρκία. Πρέπει να πω ότι και εμείς, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, Έχω να επισημάνω στον τομέα της δημοκρατίας ότι το Κοινοβούλιο με έχει απογοητεύσει πολλά πράγματα στη στάση του σε σχέση με τα προβλήματα που εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο. Και δεν θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Φιούλη. Με, τις, ε, με την Αίγυπτο καταρχάς και τις εκλογές που έγιναν πέρσι, δημοκρατικές εκλογές που εξέλεξαν τον Μούρση, ο οποίος όμως ανετράπη με ένα πραξικόπημα σήμανε και περιορισμό των ελευθεριών, της δημοκρατικής ελευθερίας έκφρασης, που συνεχίζεται εδώ και ένα χρόνο, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, ενώ ξεκινούν οι προσπάθειες για να, εντατικο... για να εδραιωθεί η δημοκρατία, η Αίγυπτος ε, παραμένει στο περιθώριο, παραγνωρίζονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Βλέπετε ότι υπάρχει μία ε, κλίμακα αξιών η οποία αλλάζει ανάλογα με την χώρα αποδέκτη ή ε, ενδεχομένω έχει αυτό να κάνει με το εάν είναι μουσουλμανικό ένα κράτος ή όχι. Η Μιανμάρ, μιανμαρ βιρμανια που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σας έχει απασχολήσει με την Αν Σαν Σουκί και τον αγώνα της για τη δημοκρατία. Έχετε βραβεύσει την Αν Σαν με το βραβείο Ζαχάροφ αλλά τον Μούρση και τον αγώνα του για την Αίγυπτο δεν τον έχετε αναγνωρίσει. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν ισχύουν τα ίδια πράγματα ή όχι. Δεν έχει την ίδια αξία η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια στην Αίγυπτο δεν έχει η ανθρωπιά τη θέση της εκεί ή μήπως είναι μόνο λέξεις. Φαντάζομαι ότι μια μέρα η Αίγυπτος θα απελευθερωθεί, θα βρει τη θέση της στο κράτος δικαίου και στην κοινωνία των ελευθέρων εθνών. Ερωτώ όμως το εξή. Όταν έρθει η ώρα και απελευθερωθεί η Αίγυπτος και είναι ελεύθερη, εσείς τότε πώς θα μπορέσετε να κοιτάξετε στα μάτια αυτών των ελεύθερων παιδιών της Αιγύπτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, τον κύριο Σαχίν. Ο κύριος Ντάφα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που θα απογοητεύσω τον κύριο Σάχιν, αλλά είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να ε, διαπιστώσουμε με πολύ ε, ε δυσαρέσκεια την την κατάσταση στην Τουρκία. Σε, σε δήλωσή σας ε, στις 3 Απριλίου με κατηγορήσατε ότι με εξαγόρασε το, το κίνημα Γκουλέν. και με αναγκάσατε να κατακρίνω την Τουρκία και να πω ορισμένα πράγματα αρκετά επικριτικά, όπως και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αυτή τη στιγμή, αδυνατεί να σεβαστεί να σεβαστεί, να εξακολουθήσει να σέβεται τα κριτήρια της Κοπενχάγης. και θα ήθελα να αιτιολογήσετε αυτές τις ε, κατηγορίες που ε, εξαπολύσατε εναντίον μου. Θεωρείτε ότι εγώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Είμαστε τμήμα αυτού που ονομάζεται μια παράλληλη δομή στην ε, Τουρκία. Και αν δεν μπορείτε να αιτιολογήσετε τις παρατηρήσεις αυτές, ε, θα ήθελα να ακούσω μια συγγνώμη εκ μέρους σας. Δύσκολα τα πράγματα. Ο κύριος Τσάνταν. Σε πολλές από τις τοποθετήσεις που ακούστηκαν νωρίτερα, στο θέμα του ανοίγματος των κεφαλαίων κτλ. Το θέμα της επανεισδοχής. Πολλά υπόθηκαν. Εκφράστηκαν θέσεις. και επικρίσεις εις βάρος της Τουρκίας. κλείστον. Έγινε λόγος για την άσκηση ε, ακραίας βίας εις βάρος των διαδηλωτών, ε, το θέμα του YouTube, του Twitter ε, και όλα αυτά. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι οι εκλογές που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζονται σε δύο θέματα, τους μετανάστες και την Τουρκία είναι όλοι κατά των μεταναστών, είναι όλοι κατά της Τουρκίας. Νομίζω ότι θα πρέπει όμως να διδαχθούμε από αυτό για να αντιληφθούμε ότι και στην Τουρκία ο εθνικισμός φέρνει ακρότητες και εντάσεις. Ίσως η Ευρώπη θα έπρεπε να κοιταχθεί στον καθρέφτη και να σκεφτεί μήπως έχει υπάρξει κάποιο λάθος από τη δική της την πλευρά και να διορθώσει την πορεία της. Ο κύριος Ερντεμίρ. Κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά είναι μια κρίση για μας, σίγουρα για την ε, τουρκική δημοκρατία, τον πλουραλισμό, την διάκριση του, των εξουσιών ε, και την ανεξαρτησία και την αμεροληψία ε, του δικαστικού τομέα. Είναι πράγματι ε, μία κρίση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα κοινά ευρωπαϊκά μας ιδεώδη, όπως επίσης και για το μέλλον μιας ε, βιώσιμης ε, ανταγωνιστικής οικονομίας. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα για μας την Τουρκία γιατί δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμη στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό με πάει πίσω σε πάνω από 60 χρόνια ε, στο στο Στρασβούργο ε, το 1949 που ο Κάσεν Λουγκέν ε, από ε, το Ρεπουμπλικανό Λαϊκό Κόμμα τότε είπε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αιώνες παράδοσης και αξιών αλλά όλα αυτά πρέπει να τα υπερβούμε και γι' αυτό είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο και ο στόχος μας πρέπει να είναι Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης. Ε, ο Άντριας Μόιτσερ, ε, ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε ότι είναι ένας συνασπισμός ε, νέγρων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όταν λοιπόν ε, αντιπαραβάλλουμε αυτές τις δύο ιδέες, δεν βλέπουμε μία αυστριακή και μία τουρκική άποψη, βλέπουμε μία ευρωπαϊκή άποψη από έναν Τούρκο βουλευτή και βλέπουμε και μία ε, ολοκληρωτική ε, άποψη την οποία εξέφρασε ένας ευρωβουλευτής. Οπότε αυτό μας ε, οδηγεί στο εξή συμπέρασμα. Δεν πρόκειται για σύγκρουση εθνών, για σύγκρουση κρατών, πρόκειται για σύγκρουση παλαιού μίσους και προκαταλήψεων, όμως εδώ είμαστε να μιλήσουμε για το μέλλον. Ένα, που ανεξα... Ένα μέλλον που ανεξαρτήτως της εθνότητάς μας και της θρησκείας Αν έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό ιδεώδες μπορούμε να το πετύχουμε. Και εμείς ε, στη μεταπολεμική Ευρώπη ε, πάντοτε είμαστε υπέρμαχοι μιας τέτοιας, ε, ενός τέτοιου ιδεώδους παρά το γεγονός ότι ευρωβουλευτές ε, ευρωβουλευτές ε, δεν ήταν πάντοτε τόσο υπέρμαχοι ενός ευρωπαϊκού ιδεόδου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνουμε μαζί, να συνεργαστούμε, γιατί ε, ό,τι θα έγιναν στην Ουκρανία δεν θα σταματήσουν εκεί, σιγά σιγά θα μας πλησιάσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα, το είπα και προηγουμένως. Ο κύριος Ραμαζάνογλου μετά ο κύριος Σογκλου και μετά θα γυρίσουμε πάλι στο βήμα. Αξιότιμη συμπρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμη πρέσβης, αξιότιμη κύριε Φίλε, Αγαπητοί συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι τη Μεγάλη Τουρκική Ευρωσυνέλευση, καλημέρα σα. Και θα ήθελα να πω ότι ζήτησα το λόγο διότι ο, η κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ, η οποία είναι και επίτροπος αρμόδια, αντιπρόεδρος μάλιστα, και επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη στις μελιώδεις ελευθερίες και την ηθαγένεια, ε, ε, έχει λάβει από πλευρά μου μια επιστολή την οποία θέλω να σας διαβάσω στα αγγλικά, γιατί είναι στα αγγλικά. Μια, ένα ανοιχτό, μια ανοιχτή επιστολή λοιπόν απευθυνόμενη στην κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ... Ευρωπαϊκή Επίτροπο για τη δικαιοσύνη στις μελιώδεις ελευθερίες και την ηθαγένεια. Αγαπητή κυρία Ρέντινγκ, είσαστε μια λαμπρή και ε, γνωστή πολιτικός του Λουξεμβούργου που έχετε υπηρετήσει σε πολλούς τομείς, εθνική και την διεθνή πολιτική ζωή. Πριν από την πολιτική σταδιοδρομία, τιμηθήκατε με τη δακτορική διατριβή σε ανθρωπιστικές επιστήμες του Πανεπιστημίου των Παρισίων της Ορβόνης, που αποτελεί μια εξαιρετική βάση για δραστηριοποίηση στην πολιτική ζωή. Στην τρίτη σας θητεία επιβεβαιώνεστε ως ε, Επίτροπος εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τη ελευθερία και την ηθαγένεια. Για να είμαστε ειλικρινεί, λοιπόν, μπορούσατε να είστε ένα πολύ καλό παράδειγμα και για πολλούς νεαρούς πολιτικούς όπως εγώ για το μέλλον. Ωστόσο δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν δέχεστε τις απαιτήσει, λέει η επιστολή, για ε, συνάντηση ραντεβού ε, που απευθύνουν σε εσά πολλοί Τούρκοι υπουργοί, παρότι σας ζητήθηκε ε, και μάλιστα σα δόθηκε ευκαιρία να προσδιορίσετε μόνοι σα την ημέρα και την ώρα τη συναντήσεω. Ποιο είναι ο σωστό δρόμο για να επικοινωνήσουμε μαζί σα, Υπάρχει ένα, ένα πρόβλημα επικοινωνία που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των προσωπικού, του προσωπικού και του γραφείου σα ή υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία για να ζητήσει κανεί ραντεβού από, από Θα ήθελα να σα παρακαλέσω να απαντήσετε στι αθώε ερωτήσει μου προσωπικά με μια επίσημη γραπτή επιστολή στην εξή διεύθυνση που παραθέτω και σας ευχαριστώ προκαταβολικά για την πολύ καλή συνεργασία και ευαισθησία που ασφαλώς θα δείξετε σε σχέση με την αιτιολογημένη και λογική διατύπωση των διπλωματικών αιτημάτων. Κυρία ε, Πρόεδρε, κυρία Φλότρο, αν μου επιτρέπετε στα γαλλικά, θα σας καταθέσω την επιστολή για να την διαβιβάσετε αρμοδίως στην κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ πολύ να κάνω και το γραμματοκομιστή. Ο κύριος Φίλε πάντως είναι συνάδελφος της κυρίας Ρέντεγκ. Ίσως είναι ο καταλληλότερος για να διαβιβάσει το αίτημα αυτό αρμοδίως. Και θα είναι και ταχύτερο. Κύριε Γκιούρ, σας ευχαριστώ. Όπως είπατε, είναι δύσκολες ημέρες. Έχουμε την κρίση της ε, Συρίας που ταρανίζει την Τουρκία εδώ και τρία και χρόνια. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδων θανάτους. Έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση μπροστά στα μάτια μας, η οποία δυστυχώς οφείλεται σε όλους μας. Όλοι μας έχουμε συνυπευθυνότητα. Έχουμε να κάνουμε με χρόνια προβλήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν. Έχουμε να κάνουμε με χρόνια προβλήματα που διωγγώθηκαν και ξεσπάνε σε μια νέα κρίση. Περάσαμε λοιπόν τη διαδικασία των εκλογών. Τοπικών και περιφερειακών εκλογών, όπου συζητήθηκε πάρα πολύ το ποιο κέρδισε και ποιο δεν κέρδισε, αλλά πάνω απ' όλα βλέπουμε ότι το θέμα είναι ότι υπάρχει ανάγκη για ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Τουρκία. ο εκλογικό μας νόμος έχει ε, καταρτιστεί κατά την περίοδο της δικτατορία του 10 Σεπτεμβρίου. Παραμένει ενισχύ. Είναι ένα νόμος δικτατορικό του εκ τούτου, ο οποίος δεν υπηρετεί τη δημοκρατία, περιορίζει πάρα πολλά δικαιώματα και ω εκ τούτου και όταν, κριθεί, η ώρα να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη δεν μπορεί να ε, γίνει ενδελεχής έλεγχος από την δικαιοσύνη. Αυτό οδηγεί σε μια πολύ βαθιά δημοκρατική κρίση. Δεν έχουμε λοιπόν διαφανεί ανοιχτέ, ανώθευτε εκλογικέ διαδικασίε. Είναι δύσκολο να πούμε κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω για άλλη μια φορά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικότερα και να καλέσω τους συναδέλφους μας όλους ιδιαίτερα για το θέμα του ανοίγματο του 23ου και 24ου κεφαλαίου. Ιδιαίτερα εμείς ως, κόμμα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας καλούμε, απευθύνουμε έκκληση θερμή να ξεκινήσει το χύτερο δυνατό η ε, διαπραγμάτευση των κεφαλαίων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουν τα κεφάλαια για τη δημοκρατία στην ε, Τουρκία. Έχουμε αντιπαραθέσεις λοιπόν Πολλέ στην Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κάποιες συγκρούσεις αιματηρές να έχουν ε, πάυσει, να έχουν διακοπεί. δεν σημαίνει αυτό ότι έχουν επιληθεί όμως τα προβλήματα. Θα ήταν μεγάλο λάθο να πιστεύει κανεί κάτι τέτοιο, γιατί το κουρδικό πρόβλημα παραμένει. Είναι ένα διεθνέ πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που αφορά τη Μέση Ανατολή ολόκληρη. Έχει να κάνει με την ε, ανθρώπινη διάσταση και το δικαίωμα στη ζωή και την ανεξάρτητη ε, ζωή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία σε επίπεδο Τουρκίας με μια ανακοχή. Μέσα στον τελευταίο χρόνο δεν έχει γίνει καμία αιματήρη σύγκρουση. Αλλά στο θέμα της επίλυσης του Κουρδικού δεν έχει γίνει και κανένα βήμα. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Ο διάλογος για να μπορέσει να οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις και συνομιλίες απαιτεί απόφαση της Βουλής χρειάζεται να προσδιοριστεί ένα πλαίσιο για τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις που να εγγυάται μια δημοκρατική, ελεύθερη ε, διαβίωση για τους Κούρδους. Εμεί πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει την υπόθεση αυτή. Αποδίδουμε πολύ μεγάλο βάρος στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως βοηθός και για τους Κούρδους αλλά και για την Τουρκία στην υπόθεση αυτή και ιδιαίτερως απευθύνουμε την έκκληση στον κύριο Φιούλε με μια ερώτηση ταυτόχρονα, σύντομη ερώτηση, εάν θεωρείτε ότι μπορεί μια δημοκρατική και πολιτική λύση να ενισχυθεί με κάποια δική σας πρωτοβουλία στο εγγύς μέλλον και τι είδους πρωτοβουλία θα μπορούσατε να αναλάβετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Για το κεφάλαιο 23 ε, θα δώσουμε το λόγο στον ε, εκπρόσωπο ε, του Συμβουλίου γιατί προφανώς θα έχει πολλά να μας πει για τα κεφάλαιο 23 και 24. Είναι κάτι το οποίο συζητούμε πολλά χρόνια και τις δικές μας απόψεις τις γνωρίζετε. Η κυρία Ιντσέκαρα. Είπατε να είμαστε σύντομοι. Θα περικόψω λοιπόν τόσο θέλω να πω. Πολύ σύντομα να σας υποβάλω τα εξή. Έχουμε γνωρίσει δυσκολίες που οφείλονται στο ότι δεν έχει μπορέσει να επιληθεί το συνταγματικό ζήτημα στην Τουρκία, παρά τις προσπαθίες μας και την βούλησή μας. Το κόμμα μας, το ΑΚΕΠΕ, έχει προσπαθήσει να ε, λύσει το πρόβλημα αυτό συστήνοντας μια, μια επιτροπή σταγματικής αναθεώρησης στην οποία ισότιμα συμμετείχαν εκπρόσωποι των εκπροσωπούμενων στην, ε, κυβέρνη, στην ε, Βουλή κομμάτων με ισότιμο αριθμό βουλευτών. Εμείς κάναμε τις προσπάθειές μας. Θα μπορούσαν ε, ακόμα, ακόμα χωρίς τη δική μας βούληση τα τρία άλλα κόμματα που συμμετέχουν στη Βουλή να συνεργαστούν και να διατυπώσουν μια αναλλακτική πρόταση συντάγματος και να την εγκρίνουν κιόλα. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Ή να εξασφαλίσουν την έγκρισή της. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτό. και βλέπουμε ότι ακόμα και η νομοθεσία η οποία στόχο έχει να διευρύνει και να ενισχύσει τα δημοκρατικά δικαιώματα μετατρέπεται σε μια ε, πηγή αντίδρασης και δυσκολιών διαρκώς. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω στον κύριο Φιούλε την εξής παρατήρηση, ότι έχουμε στην Τουρκία την, ε, το θέμα της υποκλοπής και των παρακολουθήσεων των ε, απόρριτων συνομιλιών που παρακολουθούνται παράνομα για δεκάδες χιλιάδες πολιτών της Τουρκίας και θέλω να σας ρωτήσω πώς το κρίνετε αυτό, πώς κρίνετε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των ε, δικαστικών, μεταξύ των ε, αστυνομικών, μεταξύ και των επιχειρηματιών κάποιοι οι οποίοι έχουν συνομωτήσει για να φτιάξουν μια ομάδα, μια οργάνωση η οποία ε, παρακολουθεί, υποκλέπτει συνομιλίες, ασκεί εκβιασμού Στη χώρα σας, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, πώς θα αντιδρούσατε, πώς θα το κρίνατε. Και επίσης Νομίζω ότι πολλές είναι οι προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό με πολύ καθαρό και δημοκρατικό τρόπο, αλλά όσο και αν ε, προσπαθούμε βέβαια μπορεί κάποια ε, μέτρα να χαρακτηριστούν αντιδημοκρατικά. Αλλά για το Twitter θα ήθελα να σας πω το εξή. Είπατε ότι απαγορεύτηκε κτλ. Με έχουμε να κάνουμε με επιχειρήσεις οι οποίες πολλούν υπηρεσίες και για τις οποίες, από τις οποίες η Τουρκία απέτησε να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν το πράττουν όμως. Και αυτό είναι που ζήσαμε εμείς στην Τουρκία. Έχουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα τηλεοπτικό το οποίο παρουσιάζει με μυστική κάμερα στοιχεία του απόρριτου ιδιωτικού βίου ενός πολίτου ο οποίος χωρίς να δώσει καμιά απάντηση και ε, χωρίς να κληθεί να τοποθετηθεί μέσα σε μια εβδομάδα είχε αυτοκτονήσει. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα που οδηγούν σε αύξηση των αυτοκτονιών, αύξηση της βίας, ενίσχυση της βίας κατών γυναικών, εφόσον οφείλονται στο Twitter, δεν θα πρέπει εμεί να λάβουμε μέτρα. Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ιδιωτικό βίο. Το Twitter δυστυχώ και το έχουμε δει, όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στην Ευρώπη υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Γιατί όταν είναι ανεξέλεγκτη η δράση αυτών των οργανισμών, των εταιριών κτλ., ε, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα βλέπουμε ότι η Twitter ως εταιρεία αποφασίζει να ανοίξει μια αντιπροσωπεία ε, στην ε, Τουρκία και ίσως με τον τρόπο αυτό να λυθούν τα προβλήματα. Ε, από τη Συρία επίσης. Θα ήθελα να πω ότι μπορεί να σας φαίνεται πολύ μακρινή σαν χώρα και να μην ζείτε τόσο έντονα τα δεινά και τον πόνο και τον θάνατο που αντιμετωπίζουμε εμεί καθημερινά από τη γειτονική αυτή χώρα, γιατί βλέπουμε από τα σύνορά μα το τι συμβαίνει, βλέπουμε πώ είναι οι χιλιάδε πρόσφυγες που περνούν τα σύνορα για να ζητήσουν ασφάλεια σε εμά. Δεν είναι δυνατόν όμω και εσεί να κοιμάστε ήσυχοι αν ξέρετε ότι συμβαίνουν όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να παρακαλέσουμε και μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη με μια πιο αποφασιστική δράση να πιέσετε το καθεστώς και πάνω απ' όλα να πείσετε να μείνουν τα παιδιά και οι γυναίκες εκτός αυτών των συγκρούσεων, γιατί εκεί ε, ε, εντοπίζεται η χειρότερη μορφή της σύγκρουσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φλότρο, ευχαριστώ. Ε, κυρία Τζέκαρια, ξέρετε ότι έχουμε συζητήσει το θέμα της ε, Συρίας επανειλημμένως. Δεν μπορώ να επιτρέψω να λέτε ότι οι Ευρωπαίοι είναι αδιάφοροι ή, πιο, ή δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον από ότι εσείς ε, στο θέμα της Τουρκίας. Δεν μπορείτε να μας κατηγορείτε ούτε καν για διαφορία, όσο και αν ενδεχομένω θα θέλαμε η διεθνή κοινότητα στο σύνολό τη να δείξει περισσότερη πυγμή και να είναι σε θέση να βρει μια πολιτική, βιώσιμη και διαρκή λύση στο ανθρωπιστικό, στο καταστροφικό αυτό ε, και πολύ λυπηρό ανθρωπιστικό πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ, όπως πάντα, την Τουρκία για τις προσπάθειες και το καθήκον, το βάρος που αναλαμβάνει για να υποδεχθεί αυτούς τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μακάρτη, μετά ο κύριος Γερλίκαια και μετά νομίζω κλείνουμε τον κατάλογο των παρεμβάσεων. Σας σημειώνω και έχουμε και χρόνο αρκετό για να ακούσουμε τις ερωτήσεις. Κυρία Μακάρτη, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για το θέμα του Twitter και του YouTube κτλ. Επί 10 χρόνια είχαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα στην Ευρώπη Μπορεί ο καθένα να βγαίνει στο Facebook και το YouTube ή το Twitter και να λέει ό,τι θέλει. Το Twitter είναι ένα γεγονό του 21ου αιώνα, είναι δεδομένο του 21ου αιώνα. Η απάντηση δεν είναι η λογοκρισία. Πολλοί πολιτικοί ηγέτες αντιμετωπίζουν επικρίσεις μέσω των ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο δικός μου Πρωθυπουργό ε, υπέστη σοβαρές επικρίσεις και κριτικές, ε, δεν έκλεισε το, το σύστημα γιατί δεν είναι αυτή η λύση. Εάν κάποιος έχει πρόβλημα απευθύνεται σε έναν δικηγόρο, πηγαίνει στον πάροχο της σχετικής διαγραμμικής υπηρεσίας και ζητάει να γίνει σχετική παρέμβαση για να κατέβει η σελίδα, η προσβλητική κτλ. Αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ. Δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα να κλείνουμε ένα μέσο επικοινωνίας. Διότι αν το κάνουμε αυτό, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να μειώσουμε την εμπιστοσύνη στην δημοκρατική διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως τους ε, Τούρκους συναδέλφους για το θέμα των ιδίων συμφερόντων κάτι. Ξέρετε ότι έχω, ότι έχω διατελέσει αντιπρόεδρος της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής εδώ τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχουμε μια σοβαρή οικονομική κρίση, η οποία πιστεύω και εσάς ενδεχομένως μπορεί να ρίξει σε μια σοβαρή οικονομική κρίση. Μέχρι να εμφανιστεί αυτή η πολιτική αστάθεια λοιπόν, η Τουρκία και οικονομικά πήγαινε πολύ καλά. Είχατε πολλούς επενδυτές, είχατε πολύ καλή κίνηση κεφαλαίων Τώρα όμως χαρακτηρίζεται η πιο ευάλωτη αναδυόμενη οικονομία, έχετε δυναμικό αναπτυξιακό αλλά τεράστιο εξωτερικό χρέος και εάν μειωθούν οι επενδύσεις, η εμπιστοσύνη τελικά στην οικονομία σας από πλευρά των επενδυτών, πώς θα τα βγάλετε πέρα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι κινδυνεύετε να πέστε σε μια τεράστιων διαστάσεων οικονομική κρίση όπως αυτή που αντιμετώπισε το 97 και το 1998 η Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν ως ίδιων συμφέρον να αναζητήσετε, να βρείτε λύσεις στα πολιτικά ζητήματα και την αστάθεια. Η δάτολος κινδυνεύεται με σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, μεγάλη οικονομική κρίση, ανατροπή της, ε, δυνατό, του δυναμικού ανάπτυξης που έχετε μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένας τεράστιος κίνδυνος. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι συμπρόεδροι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα και εγώ να απευθυνθώ σε εσά για να αναφερθώ στο θέμα της ελευθερίας της έκφρασης. Όπως είπε και η προλαλή σας, το κλείσιμο του Twitter ε, πώς γίνεται, γίνεται με απόφαση δικαστηρίου. Ε, μα εξήγησε ο κύριος Υπουργός ότι ε, επειδή δεν εφαρμόστηκε η δικαστική απόφαση, χρειάστηκε να ληφθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση. Αυτό ήθελα να καταστήσω πολύ το σαφές και να πω επίσης ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των τηλεπικοινωνιών στην Τουρκία βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, διότι ε, την, ε, την ουσία αυτών των δύο ελευθεριών την εξασφαλίζει η ο πλουραλισμός τα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουμε στην Τουρκία, είτε ως προς το τηλεοπτικό στο τηλεοπτικό επίπεδο τα τηλεοπτικά κανάλια. Είτε πρόκειται για ραδιοφωνικού σταθμού, είτε πρόκειται για πάρα πολλέ δυνατότητε ανάπτυξη ιστοσελίδων και ιστοτόπων μέσω του διαδικτύου. Έχουμε τα τελευταία δέκα χρόνια τεράστια προόδο και στο τεχνικό επίπεδο βεβαίω, με την ευρυζωνική τεχνολογία που έχει προωθήσει η κυβέρνηση με τι οπτικέ σύνε. Ε, υπάρχει δυνατότητα πλουραλιστικά ο καθένα να εκφράσει τι θέσει του. Στην Τουρκία έχουμε 305 εφημερίδες, των οποίων 200 περίπου είναι ημερήσιες. 700 700 τηλεοπτικούς σταθμούς, είτε πρόκειται για εθνικούς, είτε πρόκειται για περιφερειακούς, τοπικούς, τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ε, διαδικτυακή τηλεόραση επίσης πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο πλουραλισμός λοιπόν εξασφαλίζει την ελευθερία της ε, Ενημέρωση, τη έκφραση και των τηλεπικοινωνιών. Εδώ και στου τομείς αυτούς που αναφέρθηκαν μπορεί ο καθένας να εκφράσει τις θέσεις του, τις γνώμες του όπως το θεωρεί σκόπιμο. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Είναι λάθος να πιστεύετε ότι υπάρχουν εμπόδια στην έκφραση και την ε, επικοινωνία στην Τουρκία. Το θέμα του Twitter έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι μία ε, διεθνούς εμβέλειας μια μεγάλη διεθνής εταιρεία αρνήθηκε να εφαρμόσει δικαστική απόφαση. Και έτσι χρειάστηκε να παρέμβουμε. Έτσι η κυβέρνηση να παρέμβει προκειμένου να διαφυλάξει τα ε, δικαιώματα των ιδιωτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Λιγάκι ανησυχώ γιατί τα επιχειρήματα που ακούω ε, δεν μου φαίνονται πολύ αξιόπιστα. Και ανησυχώ γιατί, γιατί εμείς ε, εδώ στην Επιτροπή μας συνήθως έχουμε ειλικρινή διάλογο για ζητήματα που μας ανησυχούν για να συζητήσουμε πραγματικά και να μπορούμε να βρούμε λύσεις. Όταν προσπαθείτε να μας πείσετε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ελευθερίας έκφρασης αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, ο κύριος, ε, στην Τουρκία σήμερα, ο κύριος Παλαισάν δεν είναι εδώ, αλλά ήταν εδώ στην αρχή ε, της... Ε, ε συνεδρίασής μας και είναι ο υπεύθυνο επιτροπη Ad Hoc ε, για τη δημοσιογραφία. θα του σηκώνονταν όρθια τα μαλλιά αν άκουγαν αυτά τα πράγματα. Ε, ο Πρωθυπουργός ε, μιλά ε, με πολύ έντονο και άσχημο τρόπο κάθε μέρα για τους δημοσιογράφους. Πραγματικά Ελπίζω να ανησυχείτε κι εσείς ε, όσο και εμείς. Ελπίζω να ανησυχείτε κι εσείς για την ελευθερία έκφραση στην Τουρκία όσο ανησυχούμε κι εμείς. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια οπισθοχώρηση στην ποιότητα του διαλόγου μας. Και πραγματικά με ενοχλεί αυτό το πράγμα ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε πραγματικά και ειλικρινά για το τι συμβαίνει. Υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα τη δουλειά των δημοσιογράφων, των συνθήκων ε, υπό τι οποίε ασκούν το επαγγελμά του, την ελευθερία τη έκφραση. Ε, υπάρχουν δημοσιογράφοι ε, που είτε αναγκάστηκαν να αφήσουν το αξίωμά του με πολύ βίαιο τρόπο, είτε είναι στη φυλακή. Δεν είναι δυνατόν να μη μα ανησυχεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να διατηρήσω καν την ηρεμία μου όταν σα τα λέω αυτά τα πράγματα. Η δημοκρατία, η ελευθερία τη είναι ένας πυλώνας ε, της ε, ε, δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Δεν χρειάζεται να σας τα ξαναλέω αυτά τα πράγματα. Δεν θα ολοκληρώσουμε αυτήν την τελευταία μας συνεδρίαση στο πλαίσιο αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας υπαναχωρώντας ε, για πράγματα τα οποία αποτελούσαν και εκτιμένο όλων μας. Ε, εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσει αυτός ο πυλώνας του κράτους δικαίου. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και πολύ δύσκολες οι συζητήσεις αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε από αυτού του βασικού πράγματος. Αγαπητή εδώ βλέπουμε ακριβώς το πρόβλημα. Οι συνάδελφοι εξηγούν ότι ό,τι συνέβη στην Τουρκία γίνεται με μια προσπάθεια εδραίωση πάνω στην νομοθεσία, αλλά δεν μας ακούτε. Δεν θέλετε να μας ακούσετε και δεν θέλετε να δείτε ή να κατανοήσετε την αλήθεια. Εάν πράγματι θέλουμε να έχουμε διάλογο, πρέπει να ακούμε και ο ένας τον άλλον. Γιατί ούτε θα περνούσαν τότε κάποια θέματα που μπήκαν μέσα στην έκθεση προόδου, ούτε θα ακούγονταν κάποιες τοποθετήσεις όπως αυτές που ακούθηκαν τώρα. Εάν μονομερός γίνεται παραπληροφόρηση βάρος Τουρκίας και λασπολογία, τότε προφανώς και εσείς το εκφράζετε με τα όσα είπατε, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι αλλιώς η κατάσταση στην Τουρκία. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε με ανοιχτό πνεύμα την αλήθεια. Και τότε νομίζω κάποια από τα ε, ζητήματα που προκύπτουν και οι κατηγορίες που ακούμε να εκφράζεται δεν θα είχαν βάση και δεν θα διατυπώνονταν και θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με ένα καλό και ειλικρινή διάλογο. Τα είπαμε ε, όλα αυτά για να σας εξηγήσουμε ότι αυτά τα οποία λέτε δεν έχουν βάση. Ως Προεδρείο έχουμε λάβει μια απόφαση να μην κάνουμε σχόλια στα όσα λέγονται από τους συναδέλφους, ως πρόεδρο, πρόεδροι, συμπρόεδροι. Βλέπω ότι εσείς δεν το τηρείτε. Λυπούμε πολύ, διότι έχουμε συμφωνήσει ως Προεδρείο να απέχουμε από σχόλια. Ο κύριος Φίλε, ο κύριος Υπουργός, ο Προεδρεύων είναι εδώ παρόντες, πρέπει να δώσουν τις απαντήσεις τους και νομίζω ότι ούτε εσύ αλλά ούτε και εγώ έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. συμφωνούμε ότι όλα θα επιληθούν μέσω διαλόγου. Αλλά αν θέλουμε να επιλύσουμε κάτι, πρέπει να έχουμε κάποιο θέμα, ε, κάποιες ανησυχίες να επιλύσουμε, τουλάχιστον να είμαστε σύμφωνοι στο τι είναι η ανησυχία και το ποιο είναι το ζήτημα. Η κυρία Παβίνη τελευταία και μετά θα δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε και άλλο κατάλογο μιλητών. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Φλότρ. Πηγαίνουμε σε εκλογές ε, και μόλις ερχόμαστε από εκλογές. Ε, οπότε θα ήθελα καταρχάς ε, να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους ε, γιατί προσπάθησαν ε, να πούν στον κύριο Φιούλε και στην ε, Λέδη Άστον ότι χρειάζεται αποστολή παρακολούθησης πριν από τις εκλογές. Μας απασχολούσε πάρα πολύ αυτό το θέμα της νοθείας των εκλογών σε σχέση με το αποτέλεσμα αυτών. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα που είναι ιδιαίτερα Ε, σε μεθοριακή ε, πόλη την επομένη των εκλογών αναφέρθηκε ότι υπήρχε μία ψηφοφορία έξι ψήφων ε, διαφοράς για το κόμμα BDP στην πόλη Μαρτίν Και την επόμενη μέρα ακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών ε, γιατί υπήρχαν αντιρρήσεις από το ΑΚΠ. Ε, κέρδισε τελικά το ΑΚΠ τις εκλογές και αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να ξαναγίνουν εκλογές τον Ιούνιο. Εν πάση περιπτώσει οι εκλογές ακυρώθηκαν. Το ίδιο συνέβη ε, στη Γέλοβα όπου το ΤΣΕΧΑΠΕ ε, ανακοινώθηκε, ανακηρύχθηκε ε, ε, νικητής. Το ΑΚΑΠΕ δέχτηκε την ήττα του, αλλά τώρα το εκλογικό συμβούλιο θέλει να ξαναγίνουν οι εκλογές. Όσον αφορά τώρα την πρωτεύουσα, οι εκλογές πάρα πολύ υποπτές. Ο δικός μας υποψήφιος κατήγγειλε ε, κάθε πιθανότητα νοθείας, όμως ε, δεν δέχτηκε το ίδιο αποτέλεσμα όπως έγινε στην άλλη πόλη και για την Άγκυρα ε, το ΑΚΠ έγινε παράδοση ότι αν κάνουν ότι δεν ακούνε του, ποιοι είναι οι κανόνες, ε, αυτό γίνεται ο κανόνας τελικά. Οπότε η νοθεία συνεχίζεται. Ε, υπήρχε μια ψηφοφορία που αφορούσε ε, το θρησκευτικό νόμο έναντι στις σύγχρονες παραδόσεις και υπήρξαν ε, πολλά προβλήματα γιατί κάπου φάνηκε ότι θα μπορούσε ε, το σύγχρονο να κερδίσει το παραδοσιακό. Ε, δεν θα... Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να... Κατηγορήσουμε μια ύποπτη η οποία είναι υπεύθυνη για την πτώση του ηλεκτρικού ή πραγματικά την οθεία στις εκλογές. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν πάνε τόσο καλά όσο θα ήθελε το ΑΚΠ και όπως παρουσιάζεται τελικά. Φαίνεται ότι υποστηρίζουν κάποια πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα μεγάλα στην Τουρκία σε σχέση με το κράτος δικαίου. Υπάρχει το ζήτημα της διάκρισης των εξουσιών που βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βλέπουμε ότι παραβιάζονται όλο και πιο καθαρά στο τελευταίο καιρό, σε βαθμό που είναι ορατό για τους πάντες, η απουσία της ελευθεροτυπίας, η πόλωση, η μεγάλη, η απουσία πολιτικής εκπροσώπησης υπογραμμίζουν την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις προκειμένου να θεσπιστεί μια ε, πιο δημοκρατική και ουσιαστική ε, χώρα με το κράτος δικαίου. Είναι πολύτιμο για μας το να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία για τον εξυγχρονισμό. Για άλλη μια φορά και ιδιαίτερα στο θέμα αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης σαφώς υποστηρίζουν τη ζωτική ανάγκη και εδώ επανερχόμαστε στο θέμα και συμφωνούμε τελικά με την κυβέρνηση για άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24. Είναι απαραίτητο να συνεχίσει την πορεία αυτή για τον εξυγχρονισμό η Τουρκία. Και κλείνοντα με τα συμπεράσματα, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ λυπηρό το ότι υπάρχει τόσο χαμηλή συμμετοχή από πλευράς Ευρωβουλευτών στην σύνοδο αυτή. Μόλι το μάθαμε δε χθε το βράδυ και ότι ούτε ο Υπουργό Δικαιοσύνη θα έρθει από πλευρά τουρκική. Λυπούμεθα, λυπούμεθα βαθύτατα, διότι το 23ο και 24ο κεφάλαιο έπρεπε να τύχουν υπεράσπιση από τον ίδιο αρμόδιο Υπουργό και θα θέλαμε να τον δούμε να έρθει να μιλήσει. Okay, merci, Ξέρουμε εδώ και μια εβδομάδα ότι ο Υπουργό Δικαιοσύνη δεν θα ερχόταν, όμω είναι εδώ ο Υπουργό που είναι υπεύθυνο των διαπραγματεύσεων για τα ευρωπαϊκά θέματα και χαιρόμαστε όλο ιδιαίτερο. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε μετά με τον κατάλογο των ομιλητών, γιατί θα έχουμε πρόβλημα με του προσκεκλημένου μα, οπότε να δώσω το λόγο πρώτα στον Επίτροπο. Ε, θα συνεχίσουμε με τον κατάλογο των ομιλητών μετά. Κύριε Φίλε, έχετε το λόγο. Ελέν, ε, θα είχε την καλοσύνη να μου αφήσει να αρχίσω την ε, συνεδρίαση της ομιλίας σήμερα. Θα με αφήσει σε παρακαλώ να ολοκληρώσω καλύτερα, να μιλήσω τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία ε, Φλότρ. Θα ήθελα καταρχάς να απαντήσω στο κύριο Σαχίν για τη θέση του Συμβουλίου σε σχέση με τις ε, ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε πολλές χώρες. Όσον αφορά την Αίγυπτο, αγαπητέ κύριε Σαχίν, ήταν πολύ σαφές το Συμβούλιο. Δεν ε, τήρησε ε, σιγή. Μπορώ να σας στείλω μέσω της πρεσφείας σας εδώ τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αίγυπτο. Ζητούμε ελεύθερες και δίκαιες ε, εκλογές με, για περιεκτικό πολιτικό διάλογο. Δηλαδή θέλουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα πολιτικά κόμματα στο διάλογο αυτό και το ε, Συμβούλιο ε, δεν παρέμεινε σιωπηλό. Νομίζω ότι είπα ότι εκπρόσωπος σήμερα είναι στην Αίγυπτο. Εχθές ήταν στο Κάιρο, έχει πάει πολλές φορές στο Κάιρο, προσπαθώντας ε, να παροτρύνει πραγματικό πολιτικό διάλογο και ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στην Αίγυπτο. Αλλά μπορώ να σας στείλω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και μπορείτε να διαβάσετε την ε, θέση των 28 κρατών μελών. Αυτά για την Αίγυπτο. Συγγνώμη, δεν μπορώ να δεχθώ ότι το Συμβούλιο ε, παρέμεινε σιωπηλό σε σχέση με τα γεγονότα στην Αίγυπτο. Όσον αφορά τώρα το άνοιγμα περισσότερων κεφαλαίων και συγκεκριμένα των 23 και 24, εγώ ε, εκπροσωπώ το Συμβούλιο, αλλά μπορώ να σας εξασφαλίσω, δεν μπορώ να μιλήσω για κάθε κράτες μέλος ξεχωριστά, αλλά εκπροσωπώ το Συμβούλιο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει πρόοδος σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έχουν αρχίσει. Ε, όμως το άνοιγμα περαιτέρω κεφαλαίων ε, εξαρτάται από τις προσπάθειες της Τουρκίας, γιατί ο γνώμονας είναι η πρόοδος Τουρκίας σε σχέση με τα ορόσημα, όπως επίσης και η κάλυψη των όρων της ένταξης και της προσχώρησης. Ε, επίσης, εξίσου σημαντικό, το άνοιγμα των ε, οκτώ ε, κεφαλαίων εξαρτάται από την ε, εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων ε, της ε, Τουρκίας σε σχέση με τις συμφωνίες και τα πρωτόκολλα που έχει υπογράψει. Η κυρία Όμεν έχει φύγει, αλλά το είπε και εμείς ως Συμβούλιο θα συμφωνούσαμε αν η Τουρκία προέβαινε σε περισσότερες μεταρρυθμίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανεξαρτήτως του ανοίγματο των κεφαλαίων. Το ε, Συμβούλιο, η Προεδρία θα ήθελε να ανοίξουμε περισσότερα κενά κεφάλαια το συντομότερο δυνατόν, όμως οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα που ανέφερα δεν έχουν καμία σχέση με το άνοιγμα των κεφαλαίων εμείς θα επικροτούσαμε κάθε προσπάθεια και κάθε μεταρρύθμιση από την Τουρκία και από τα πολιτικά κόμματα της Τουρκίας προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, Νομίζω κύριε Πρέσβη ότι για τον ε, συνάδελφο Σαχίν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τη δήλωση της κάθε άστον, ε, την πολύ σαφή σε σχέση με ε, τις θανατικές καταδίκες στην Αίγυπτο. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη και πολύ σαφής ε, στις απαντήσεις της και στην αντίδρασή της. Από την αρχή ήταν έτσι σε σχέση με τα γεγονότα στην Αίγυπτο και σε σχέση με τον πρόεδρο Μόρση. Ξέρετε ότι πάρα πολύ σαφώς εξέφρασε την αγανάκτηση για τη θανατική καταδίκη των 500 αδελφών μουσουλμάνων στην Αίγυπτο. Το είπε σαφέστατα, κάθα, κατακάθαρα και ελπίζουμε ότι με τις πιέσεις μας και χαίρομαι που το λέτε γιατί αυτές οι πιέσεις πρέπει να είναι ε, έντονες ε, ε, θα μπορέσει ε, ο μεγάλος ο μεγάλος μουφτής θα μπορέσει να ε, ανακαλέσει την απόφασή του αυτή. Ελπίζω πάντως και είμαι βέβαιη ότι η Λέδη Άστον ε, ήταν πάρα πολύ αδιάλακτη και πάρα πολύ σαφής σε σχέση με αυτά που είπε για την ε, Αίγυπτο. Και αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τη δήλωσή της για να το διαβάσετε και ο ίδιος. Εκτός μικροφώνου η Πρόεδρος. Η θέση του Συμβουλίου ήταν πάρα πολύ σαφής ε, από την αρχή, όχι μετά τις θανατικές καταδίκες, αλλά από την αρχή. Voilà. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ε, ξέρουμε το τι έγινε στην Αίγυπτο. Ε, ήταν σαν πραξικόπημα αυτό που έγινε. Είδαμε όλα τα χαρακτηριστικά να εξελίσσονται όσο περνούσε ο καιρός.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 Υπήρχε μια πολύ σημαντική ερώτηση και από, την, ε, τον κύριο Νταφ και από την κυρία ε, Όιμεν Ρόιτεν. Ε, σας ζήτησε ο κύριος Νταφ να επεξηγήσετε αυτά που είπατε ει βάρο του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευκαιρία σας για να απαντήσετε στον πρόεδρο των πολιτικών ομάδων που σας μίλησε για την κατάσταση το, των γυναικών ε, Φυσούν Ερδογάν και Πινάρ Σελέκ είναι κάτι το οποίο μας φαίνεται πραγματικά απαράδεκτο αυτό που έγινε. Οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων σας απέστειλαν επιστολή και σας ζήτησαν να ε, σταματήσει αυτή η νομική παρενόχληση ε, ούτε για τη μία ούτε για την άλλη υπάρχει καμία απολύτως υποψία. Εδώ και 16 χρόνια η Πινάρ Σελέκ παρενοχλείται ε, όλο και περισσότερο συνεχίζεται αυτό ε, και η Φιζούν Ερντογάν ε, μετά από 7 χρόνια είναι ακόμη φυλακισμένη χωρίς καμία απόδειξη εις βάρος της. Το είπατε κιόλα. Υπάρχει αυτός ο νόμος για την παράνομη κράτηση πάνω από 5 χρόνια απαγορεύεται και είναι κρίμα όπως ε, και ε, οι δολοφόνοι ε, του η ωραία της Μαλάτια απελευθερώθηκαν, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σημερινή ευκαιρία για να μπορέσετε να απαντήσετε στο στα σχετικά ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Συμπρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στην κυρία Όμεν Ρόιτσεν για τις σκέψεις και τις ε, τοποθετήσεις της. Από αυτά που είπαμε, μάλλον κατάλαβε λάθος ή ίσως και μεταφραστήκαμε λάθος. Εγώ δεν είπα ότι δεν αναλαμβάνει βήματα μεταρρυθμίσεων η Τουρκία επειδή δεν έχουν ανοίξει κάποια κεφάλαια. Είπα αντίθετα ότι ανεξαρτήτως του αν ανοίγουν τα κεφάλαια, παρά το ότι δεν ανοίγουν τα κεφάλαια, εμείς κάνουμε τι μεταρρυθμίσει μας, έχουμε τις ομάδες εργασία, έχουμε τις επιτροπές και υποεπιτροπέ σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεχίζουμε εντατικά τις εργασίες μας, αδιάκοπα. Ε, είπαμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης για την, ε, ε, αντιμετώπιση των παραβιάσεων της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με συνεδριάσεις που γίνονται σε άτυπο επίπεδο, αλλά κάνουμε τα σχετικά βήματα, κάνουμε και τις μεταρρυθμίσεις μας όπως προβλέπεται ανεξαρτήτως του εάν ανοίγουν τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων εμείς συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό έργο. Ε, ε, το να κάνουμε εμεί προσπαθίε μα. Αλλά παρόλα αυτά να μα λέτε ε, δεν έχετε καμιά προοπτική να ανοίξουν τα κεφάλαια, πάλι μα απογοητεύει πολύ. Στο θέμα τη Κύπρου, στο, ε, στη στάση τη Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία και γενικότερα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό, αισθανόμαστε μεγάλη απογοήτευση. Δυστυχώ. Πάντω, το πλαίσιο του διαλόγου υπάρχει. Μέσα στον τελευταίο χρόνο έχει προχωρήσει. Υπάρχει μία βάση ε, και ένα θεματολόγιο με διαρκή επικοινωνία και συναντήσεις με τον κύριο Φιούλε, με το θετικό θεματολόγιο ε, και με συναντήσεις και συνομιλίες για τα διάφορα θέματα που μπορούν να μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε. Δεν μπορείτε όμως να μας κατηγορείτε ότι δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Εμείς θέλουμε πιο πολύ engagement πιο πολύ δέσμευση, πιο πολύ αποφασιστικότητα και να αναγνωρίσετε βεβαίω ότι έχουμε κάνει τα, βήματά μα, ότι έχουμε φέρει νέα πακέτα μεταρρυθμίσεων και συνεχίσουμε. Για το θέμα του κυρίου Γκύρ ότι δεν γίνονται προσπάθειε για την επίλυση του κουρδικού και των δημοκρατικών δικαιωμάτων με απογοητεύεται. Με απογοητεύεται δεν περίμενα ότι θα ακούγα κάτι τέτοιο από εσά γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κύριε Γκύρ ότι έχουμε πραγματοποιήσει πολύ σημαντικά βήματα ε, θα μπορούσατε να πείτε γίνανε βήματα αλλά δεν αρκούν. Θα το δεχόμουν. Και εγώ θα έλεγα ότι ναι, χρειάζεται να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν γίνονται βήματα. Έχουμε παραδείγματι την ε, νέα νομοθεσία η οποία επιτρέπει τη χρήση των κουρδικών ονομάτων, των κουρδικών γραμμάτων του αλφαβήτου, τη δυνατότητα για διδασκαλία τη κουρδική γλώσσα στο σχολείο. Ε, μια σειρά από δικαιώματα που αποδίδονται και αναγνωρίζονται στον κουρδικό, στους, ε, στους Κούρδους. ως εκ τούτου βλέπετε ότι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία της σκέψης είναι υπό την εγγύηση της τουρκικής, του τουρκικού κράτους ενώ στο παρελθόν ε, και μόνο η υποστήριξη ηλεκτική προς μια τρομοκρατική οργάνωση ε, θεωρούνταν ε, αδίκημα, ποινικό, τώρα μόνο η εν προσφορά υποστήριξης σε τρομοκρατικές οργανώσεις μπορεί να είναι αδίκημα. Αυτά είναι σημαντικέ αλλαγέ, είναι σημαντικέ εξελίξει. Δυστυχώ όμω και παρόλε τι προσπάθειε που έχουμε κάνει, είδαμε ότι στην προεκλογική εκστρατεία σε μεγάλο βαθμό οι Κούρδοι συνάδελφοι ε, είχαν διαφορετικές ευκαιρίες θα έλεγα σε σχέση με τους λοιπούς υποψηφίους οι οποίοι υπέστησαν ακόμη και σωματική βία και επιθέσεις. Για την κυρία Μακάρτη που είπατε ότι πρέπει να αποφασίζει κανείς να προσφύγει στο δικαστήριο εάν βλέπει να παρεμβάζουν τα δικαιώματά του από το Twitter ή κάποιο άλλο δίκτυο. Ναι, να σας πω. Για το Twitter έχουμε 400 περίπου δικαστικές αποφάσεις κατά του Twitter. Όχι που έχει προκαλέσει η κυβέρνηση, αποφάσεις που απορρέουν από κάποια προσφυγή κάποιου πολίτη, ιδιώτη. Γιατί παραβιάστηκαν τα ατομικά του δικαιώματα, οι ατομικές ελευθερίες και το δικαστήριο έχει ως εκ τούτου εκδώσει απόφαση για διακοπή ε, για, της ανάρτησης, για άρση της ανάρτησης κτλ. Καθώς όμως το Twitter ε, δεν σέβεται, γιατί όταν έρχεται η εντολή από Αμερικανικό δικαστήριο αφαιρεί τη σχετική ανάρτηση το Twitter, όταν έρχεται ε, από τη Γερμανία για θέματα ναζισμού τα, αφαιρεί επίσης, α, αφαιρεί τι αναρτήσει, το ίδιο και από τη Γαλλία για θέματα προδεξιά, Όταν όμως έχουμε εμείς η Τουρκία κάνει τέτοια κίνηση για να ζητήσουμε να αφαιρεθούν κάποιε αναρτήσει προσβλητικέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μα αγνοεί. Άρα λοιπόν πρέπει και να μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση και να ζητήσουμε την αποκατάσταση του δικαιώματο σωστά. Όπω εφαρμόζει το Twitter τι δικαστικέ αποφάσει στη δική σα στην πατρίδα, πρέπει και στην Τουρκία. Έτσι δεν είναι. Εάν βγει μια δικαστική απόφαση ενός, ε, κατά ενό ε, τηλεοπτικού σταθμού στην Αγγλία, δεν θα την ε, ακολουθήσει, δεν θα υποταχθεί στην ετοιμιγορία της. Ε, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα μέσα δικτύωσης, με τα μέσα του ίντερνετ. Και στη δική σας πατρίδα όπως και στη δική μου. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόζονται δικαστικές αποφάσεις και να τη χάνουν σεβασμού από τον καθένα. Η ε, κρατική εξουσία προέρχεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκφράζεται μέσω της δικαστικής αποφάσεως και αυτή πρέπει να υλοποιείται. Αυτά είχα να πω για την αγαπητή συνάδελφο. Για δε τις εκλογές, Όντω, ανέβηκαν πολύ τόνοι στην προεκλογική περίοδο. Άμα κοιτάξουμε βέβαια τι ευρωεκλογέ και την, την πορεία ενόψη των ευρωεκλογών, και εκεί πέρα βλέπουμε ότι ανεβαίνουν οι τόνοι, εμφανίζεται ο ρατσισμό, εμφανίζεται ο αντισλαμισμό, η ξενοφοβία. Ε, προσπαθούν κάποιοι να κερδίσουν ψήφου με τον τρόπο αυτό. Λυπούμαστε πάρα πολύ βέβαια. Τα πολιτικά κόμματα και οι υποψηφοί του θα ήταν καλό να κοιτάξουν να λύσουν τα εσωτερικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμεριστούν με τους ψηφοφόρους τους λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Ίσως τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λιώνονταν με μια πιο ε, δυναμική πολιτική διεύρυνση, επί παραδείγματι. Αλλά αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί. Κοιτάξτε να σα πω πάντω, ε, ό,τι, και, ό,τι να εκφράστηκαν από ορισμένα κόμματα δεν επηρέασαν την εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία. Έδωσαν την ψήφο του οι πολίτε, έδωσαν την ψήφο του στην οικονομική ανάπτυξη. Έδωσαν την ψήφο του στο κόμμα που εργάζεται για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοκρατία στην, στην ε, Τουρκία. και ήταν πολύ οι ψηφοφόροι, παλαιοί ψηφοφόροι του δεύτερου κόμματο τη αντιπολίτευση, τη ίσονο αντιπολίτευση όπω λέμε, του ΜΕΧΕΠΕ δηλαδή, που έδωσαν την ψήφο του τελικά στο ΑΚΠ. Ε, μετά λοιπόν τις εκλογές αυτές βλέπουμε ότι ενισχύεται η αξιολόγηση της Τουρκίας ως ε, χώρου επενδύσεων. Έχουμε πολύ θετικές αξιολογήσεις. Το Μάρτιο η ανάπτυξη των ε, εξαγωγών παρουσιάζει έως και 4% αύξηση. Έχουμε δυναμικό ανάπτυξη πολύ μεγάλο, το χρηματιστήριο παρουσιάζει σημαντική άνοδο επίσης και τα επιτόκια πέφτουν σε μονάδες πλέον, εκφράζονται πλέον σε μονάδες. Η παραγωγικότητα δε και το δυναμικό παραγωγής Τουρκίας όλο και ενισχύεται. Οπουδήποτε και αν κοιτάξουμε τα οικονομικά ζητήματα μπορεί για κάποια πολιτικά να παραμένουν κάποια ερωτηματικά, αλλά στα οικονομικά ζητήματα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχία, δεν υπάρχει κανένα πεδίο αστάθεια ή αποσταθεροποίηση. Είναι βεβαίω πρώτα απ' όλα κύριος στόχος μας η πολιτική σταθερότητα. Ε, για την κυρία Παβέη. Μιλήσατε για την, ε, την Σαρία και ότι κινδύνεψε η Τουρκία να πέσει στα χέρια της, ε, των υποστηρικτών της Σαρίας. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που είπατε. Δεν υπήρξε το θέμα ποτέ στην Τουρκία. Ε, απλώς κάποιοι προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν και να παρουσιάσουν τέτοιου είδους εικόνα στην προεκλογική τους εκστρατεία. Εμείς έχουμε να κάνουμε με επιλογή ανάμεσα σε καλούς δημάρχους και κακού δημάρχου. Δημάρχου που είχαν να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την πόλη του και έργα και άλλου που δεν είχαν σχέδιο. Είδατε ότι γίνανε ενστάσει για τη Γιάλοβα, έγιναν οι ενστάσει και κέρδισε τελικά το JHP με μικρή διαφορά. Δεν είπατε όμω το εξή, ότι και οι δύο υποψήφοι και του Μπέντεπε στο Μάρτιν και του ΑΚΕΠΕ συνεννοήθηκαν και ζήτησαν από κοινού την επανάληψη των εκλογών στο Μάρτιν. Αυτό ξεχάσετε να το πείτε και δίνετε λάθος εντύπωση. Συμφώνησαν τα δύο κόμματα και είπαν ότι πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Έτσι η η απόφαση για επανάληψη της ψηφοφορίας. Είναι συνενετική, γιατί ήταν πολύ σημαντική η ψηφοφορία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως θα βοηθούσε να αποδείξει πόσο λογικά και ψύχραμα έγινε η εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία. Για τα άδανα που έγιναν πάλι ενστάσεις την ένσταση την έκανε το κόμμα της κυρίας Παβέη. Καταχρηστικά. Το δε ανώτατο εκλογικό συμβούλιο έκανε μία πολύ σημαντική αλλαγή αυτή τη φορά με την ταχύτατη επεξεργασία των ενστάσεων μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Από την ώρα που διατυπώθηκε η ένσταση, αμέσως προέκυψε η επεξεργασία των ε, ενστάσεων. Και στο Σαριέρ και στο Εσκίσεχυρ που γίνανε αντίστοιχες ενστάσεις, τις δέχθηκε και έκανε την επανακαταμέτρηση. Στο Εσκίσεχυρ, παραδείγματι, κέρδισε το GHP ε, για άλλο κοιτάξτε, δεν υπάρχει θέμα ακύρωση ή ακυρότητα. Υπάρχει ζήτημα μόνο διερεύνηση του αν αυτοί που ψήφισαν ήταν και εγγεγραμμένοι στους, ψηφ... στους καταλόγους των ψηφοφόρων. Είχαν δικαίωμα του εκλέγην δηλαδή. Δεν ήταν ζήτημα δηλαδή απάτηση ή νοθείας ως προς την καταμέτρηση των ψήφων. Ήταν κάτι που είχε να κάνει με την επαλήθευση των εκλογικών καταλόγων. Επίσης για την Πινάρ Σελέκ και την Φουζούν Ερντογάν. Δικαστικές αποφάσεις. Ε, είναι ένα θέμα της δικαιοσύνης. Ξέρετε ότι η Πινάρ Σελέκ ε, με μια κατηγορία ότι έχει εμπλακεί σε τρομοκρατική επίθεση με βόμβα στην ε, Κωνσταντινούπολη έχει καταδικαστεί. Ακυρώθηκε η καταδίκη της από, από ανώτερο δικαστήριο, ανώτερο δικαστήριο. Η Φουσούν Ερντογάν έχει απαλλαγή από, την, από το δικαστήριο για την οποία απαλλακτική απόφαση εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλιο, μπορούμε να πούμε βέβαια αν είναι δίκαιη ή άδικη αυτή η απόφαση και να διεκδικήσουμε να ε, ξαναγίνει η αξιολόγηση. Για την Πινάρ Σελέκ ε, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εμένα με ενδιαφέρει να δω αν υπάρχουν βάσιμα αποδεικτικά στοιχεία που προσφέρονται στην ε, δικαστική κρίση και που μπορούν να πείσουν το δικαστήριο. Γιατί φουζούν Ερντογάν ε, που απαλλάχθηκε από την κατηγορία της συμμετοχής και μάλιστα της ηγεσία σε ε, τρομοκρατική οργάνωση, αυτά είχα να πω. Για την ε, περίπτωση δε των φερωμένων ως δολοφόνων του ιερέως της Μαλάτια ή άλλων πιθανών ε, εγκληματιών ή τρομοκρατών, ε, αυτοί δεν έχουν ε, απαλλακτική απόφαση λάβει. Άρα ισχύει ο νόμος ο σχετικός με την προσωρινή κράτηση, εφόσον τα δικαστήρια δεν έχουν μπορέσει μέσα στην πενταετία να εκδώσουν απόφαση, πρέπει να παρέμβει η νομοθεσία. Αυτά δυστυχώ, βλέπουμε να παραμένουν ω παρακαταθήκη του παρελθόντος, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και τώρα θα ήθελα να πάτσω στον κύριο Νταφ για την ερώτησή του. Αγαπητοί φίλοι, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Εγώ πρέπει να ξέρετε ποτέ δεν θα έκανα τέτοιου είδου δηλώσει. Αλλά όποιο σα μετέφερε αυτά τα λόγια μου, θα ήθελα να σα πω ότι σα κορόιδεψε, σα είπε ψέματα. Εμένα δεν είναι δυνατόν από το στόμα μου να βγουν τέτοια λόγια, όπω αυτά που μου αποδίδεται. Δυστυχώς μόνο στα αγγλικά ακούστηκε, στις αγγλικές ειδήσει ακούστηκε με τέτοια διατύπωση. Στις τα ειδήσει τέτοιου ίδιου πράγμα δεν υπάρχει. Η ερώτηση που μου είχε απευθυνθεί ήταν η εξή. Ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση πολιτική ως προς την εξουσία στην Τουρκία και η δυνατότητα της πολιτικής, ε, μιας παράλληλης πολιτικής δομής. Και με ρωτήσανε εάν ε, υπάρχει περίπτωση, όπως λένε οι New York Times, να επηρεάσει αυτό τη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λοιπόν απάντησα ότι ένας φιλελεύθερος βουλευτής, ο κύριος Δαφ, μπορεί να σκέφτεται κάτι τέτοιο και σεβόμαστε τις θέσεις του, γιατί είχατε κάνει μια ε, πρώτος ψηφίσματος στην Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων, ε, για την οποία δεν, ε, η οποία πρότεινε να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις και για την οποία δεν είχατε την υποστήριξη των συναδέλφων σας. Δεν είναι κρίθη από τους λοιπούς. Βλέπω λοιπόν ότι οι απόψεις ενός Ευρωβουλευτού και μόνο, η δική σας δηλαδή πρόταση να διακοπούν αυτές ε, διαπραγματεύσεις ε, δεν ε, μετατράπει σε απόφαση των 776 βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. έτσι λοιπόν, καλό θα είναι να μην μεταφέρονται αυτά, αυτές οι ειδήσει σαν να σκοπεύει, στην τουρκική κοινή γνώμη πλέον, σαν να σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Γιατί μια τέτοια απόφαση, η οποία μάλιστα δεν πέρασε καν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μπορεί ούτε να δεσμεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε να έχει ε, αντίκτυπο στη σχέση με την της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δεσμεύει την τουρκική κυβέρνηση. Το να μεταφέρονται από τους New York Times ειδήσει που έχουν να κάνουν με την προσωπική άποψη ενός Ευρωβουλευτή μεμονωμένου και να παρουσιάζονται ως συνολική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αντίκτυπο στην τουρκική δημοκρατία δεν μπορεί να είναι σωστό. Αυτό είπα. Δεν σας κατηγόρησα για τίποτα. Είπα ότι είστε μεμονωμένος ο Ευρωβουλευτής και εδώ βλέπω ότι και εσφαλμένα παρουσιάζεται η κατάσταση και ε, εμφανίζεται μία μεμονωμένη τοποθέτηση ως εσφαλμένα όσο... Ε, ε, απόφαση που εκφράζει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα στον δημοσιογράφο, ούτε εσεί φταίτε γι' αυτό, ούτε εγώ φταίω γι' αυτό, αλλά πρέπει κάπω να αλλάξει και να, η κατάσταση και να μην μεταφέρονται ψευδεί ειδήσει. Αυτό είπα μόνο. Merci, Monsieur le Ministre. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τις ε, απαντήσεις σας που ήταν ειλικρινείς, ε, διεξοδικές ε, και πολύ ακριβείς, πολύ συγκεκριμένες. Ο Επίτροπος Φίλε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν ε, μιλούσαμε για την ενίσχυση της ε, δημοκρατίας ε, στην Τουρκία και εμέσως συνεχίζω αυτά που υπόθηκαν πριν από λίγο, Πάντοτε μας έκαναν εντύπωση τα δύο επιπρόσθετα στοιχεία στην Τουρκία που έπαιζαν έναν σημαντικό ρόλο. Το πρώτο ήταν η ύπαρξη των ε, θεωριών συνωμοσίας ως ε, ε, λόγων για όλες αυτές τις δυσκολίες και μερικές φορές αυτό το καθιστούσε πολύ πιο εύκολο για τις αρχές να αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα αποφεύγοντας τους πραγματικούς λόγους πίσω από αυτές τις δυσκολίες. Δεύτερον, ήταν οι εκλογές ε, που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να διαλέξει ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Όμως με τα... μερικές φορές ξεχνάμε ότι για να λειτουργήσουν αυτές οι εκλογές ως τέτοιες πρέπει να υπάρχουν οι σωστοί θεσμοί από πίσω, τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν ε, στους ε, ανθρώπους που θα εκλεγούν να ε, επιτύχουν όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκαν στην προεκλογική περίοδο μάλιστα με δημοκρατικό, περιεκτικό και διαφανή τρόπο. Κάτι ακόμη θα ήθελα να πω μετά από αυτή την ε, γενική παρατήρηση για τις εκλογές. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι ότι οι ισχυρισμοί ε, παρατυπιών πρέπει να παρακολουθηθούν με διαφανή τρόπο και πλήρως. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί το αποτέλεσμα των εκλογών δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια αμφιβολιών, γιατί είναι ο μόνος τρόπος, η μόνη βάση αποδοχής των αποτελεσμάτων των εκλογών από όλους και στην προκειμένη περίπτωση από όλους, ε, όλα τα ε, τουρκικά κόμματα και από όλους τους ε, πολίτες. Τώρα, όσον αφορά την ξενοφοβία και τον λαϊκισμό, μας απασχολεί αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά και μας απασχολεί. Κατά πόσο το εκφράζουμε, βεβαίως και το εκφράζουμε. Ψάχνουμε δικαιολογίες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, αυτό φυσικά και όχι, γιατί δεν υπάρχουν θεωρίες ε, ε, συνωμοσία πίσω από όλα αυτά. Μόνο τα δικά μας λάθη και οι δικές μας αδυναμίες. Με απασχολεί όμως και το εξής ότι αυτή η αυξανόμενη τάση ε, λαϊκισμού λαμβάνει χώρα τη στιγμή που μια σημαντική ευρωπαϊκή χώρα αποφάσισε να αγνοήσει ε, την ε, πράξη του Ελσίνγκη του 1975 και να θέσει τους δικούς της κανόνες για ε, την Ευρώπη. Αυτό όχι μόνο μου δημιουργεί ανησυχία, αλλά μου δημιουργεί και τρομερή αμηχανία. Και αυτό εξηγεί πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε αυτήν την μοναδική στρατηγική μας σχέση με την Τουρκία. Γιατί κανένας από μας ε, δεν θα έβγαινε κερδισμένος ε, εάν αυτές οι δύο τάσεις που ανέφερα ε, ενισχύσουν η μία την άλλη. Τρίτον, το κουρδικό ζήτημα. Έχουμε πολλές φορές ε, εξηγήσει πόσο ε, σημαντική είναι αυτή η ειρηνευτική διαδικασία που ξεκίνησε το 2013 και ποτέ δεν ε, σταματήσαμε να το τονίζουμε αυτό και να λέμε ότι είναι προσώφη. Όμως, πέρα από αυτό αυτή την πολιτική διάσταση, υπάρχει και μία ακόμη διάσταση. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι οι μεταρρυθμίσεις ε, για την, ε, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ε, έκφρασης και για το κράτος δικαίου, δημιουργούν πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες για την αντιμετώπιση των ε, ε, ζητημάτων αυτών. Και το τρίτο θέμα, σε σχέση με το κουρδικό ε, ζήτημα, και θα ήθελα να το επανυπεβεβαιώσω αυτό, είναι ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και μέσω ε, προενταξιακής ε, ενίσχυσης. ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η λύση θα είναι επικερδής ε, για όλους τους Κούρδους. Κάτι ακόμη, επαναλαμβάνω τώρα αυτό που είπε η Ελένη για την ελευθερία της έκφρασης, Ο αριθμός ε, των ε, εφημερίδων δεν είναι βασικό επιχείρημα υπέρ της ελευθερίας ε, του λόγου και της ελευθερίας έκφρασης. Και το να λέμε επίσης ότι υπάρχει νομοθεσία και ότι είναι τέλεια, που δεν είναι βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι εφαρμόζεται σωστά. Οπότε πραγματικά Αναμένω εναγωνίως το Μάιο την αξιολόγηση ομοτήμων που θα επικεντρωθεί κυρίως σε αυτό το θέμα και τότε θα δουλέψω και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Τουρκικό ε, Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί η έκθεση να φανερώσει. Το πέμπτο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι κρίσιμο. Μπορεί κάποιοι να το θυμάστε, το είπα αυτό και κατά τις ακροάσεις, είχα πει ότι νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας και από τις δύο πλευρές και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από την πλευρά της Τουρκίας. Και τότε είχα πει σαφέστατα ότι όσον αφορά την αξιοπιστία της Τουρκίας ότι συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει. Το κάνει επιλεκτικά και το είχα πει αυτό, ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, είναι ε, ο μοχλός, ο κινητήριος μοχλός ε, των, της διαδικασίας προσχώρησης και είχα επίσης καταστήσει σαφές ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Οι πολιτικοί αμφισβητούν ε, τον τελικό στόχο της διαδικασίας προσχώρησης. Αυτό δεν είναι και αυτό πρόβλημα αξιοπιστίας. Θα λέγα πως ναι. Επιπλέον, κάποια κράτη-μέλη που δεν μας επιτρέπουν ε, να ε, χρησιμοποιήσουμε πλήρως ε, τις δυνατότητες ανοίγματο και άλλων κεφαλαίων και αυτό δεν είναι πρόβλημα αξιοπιστίας. Ναι, είναι πρόβλημα αξιοπιστίας. Εντάξει, είναι σαφή τα ορόσημα ότι χρειάζεται να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα κρίνουν την απόδοση σε σχέση με αυτά τα ορόσημα το να γίνει αυτό λογικά θα πρέπει να σημαίνει ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Με ρωτήσατε πώς είναι δυνατόν ε, να ε, μην μπορείτε να δεχθείτε τα αποτελέσματα των επιδόσεων ε, στην, στα, στα ορόσημα αυτά. Και είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να το κάνει αυτό επί συγκεκριμένων ζητημάτων και δεν μπορώ να, να καταλάβω πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι αυτό είναι ε, προς συμφέρον είτε της Τουρκίας είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δουλεύουμε πολύ σκληρά για το άνοιγμα του κεφαλαίου 23 και του 24 και αν δει κανείς το θέμα, το σχέδιο δράσης ε, και το διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και το τι θα κάνουμε εκεί, θα ασχοληθούμε με πολλά από αυτά τα θέματα που ανήκουν σε αυτά τα δύο κεφάλαια. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε, όμως αναρωτιέμαι το θετικό πρόγραμμα δεν στερείται νοήματος. Όντως κάναμε πολλά πράγματα. Ιδρύσαμε ομάδες εργασίας με την υποστήριξη ε, του Συμβουλίου για τα ε, κεφάλαια ε, για τα κεφάλαια Αν όμως με ρωτήσετε πόσες φορές αυτή η ομάδα εργασίας για το κεφάλαιο 23 συνήλθε πέρσι ή φέτος, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να απαντήσω. Καμία φορά. Και όταν λέω ότι χρειαζόμαστε μία νέα, μία ανανεωμένη δέσμευση, μιλάω για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα έπρεπε και οι δύο να εποφεληθούμε προσπαθώντας να ανοίξουμε επισήμως το κεφάλαιο 23 γιατί επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι είναι προ συμφέρον και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Τουρκία. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που υπάρχει ήδη αντί να αναζητούμε δικαιολογίε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, σαφέστατα, ότι είμαι όσο πιο ευέλικτος και όσο πιο ρεαλιστής μπορώ να είμαι, ε, στο να βοηθήσω τις τουρκικές αρχές να αξιοποιήσουν το δυναμικό ε, που υπάρχει για το άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών, για όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα. Και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω αφορά το εξής. Εγώ περιμένω ε, έναν ανοιχτό, ε, επικοδομητικό, ειλικρινή ε, διάλογο μαζί σας. Δεν θέλω μόνο να ανταλλάσσουμε απόψεις λέγοντας ότι υπάρχει απογοήτευση και υπάρχει απογοήτευση και από τις δύο πλευρές, όμως πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να χειριστούμε την περίοδο τη χρονική από τώρα μέχρι την έκθεση προόδου. Γιατί θα ήθελα η έκθεση προόδου του 2014 να δείξει περισσότερη πρόοδο σε σχέση με αυτή του 2013. Και δεν έχουμε καταφέρει κάτι τέτοιο για την ώρα. Πρέπει πραγματικά να δουλέψουμε πολύ σκληρά, να βάλουμε τάξη και οι δύο, ε, και η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες των πολιτών μας. Κάτι ακόμη. Το πόσο περιεκτική θα είναι όλη η διαδικασία. Είναι για μένα εξαιρετική σημασίας εκτός από τους, τις συνομιλίες ε, με τον Αχμέτ Νταβούτογλου, ε, με τον Πρωθυπουργό, ε, να υπάρχει και ένας ειλικρινής διάλογος σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Η Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό. Ε, μια Τουρκία με μια ζωτική ε, κοινωνία των πολιτών πρέπει να επωφεληθεί από αυτά για τα οποία συζητούμε και για τις διαδικασίες, ε, από τις διαδικασίες ε, για τις οποίες προσπαθούμε να αποφασίσουμε, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να αποφύγουμε την ε, διωγγούμενη πόλωση εμείς δεν είμαστε εδώ για να σας επιβάλλουμε κανένα μοντέλο για το πώς θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα αυτά. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, να σας, προσφέρουμε ένα, να σας προσφέρουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, για να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση προκειμένου η Τουρκία να μπορέσει να ε, επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Και δεν ε, και να μην ε, τα καλύψει, να μην τα κρύψει απλώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε Φούλε. Νομίζω ότι καταδείξατε αν χρειαζόταν ε, αν τα ωφέλη όλης αυτής της διαδικασίας ε, και μας δείξατε και πόσα πολλά κάνατε εσείς ε, με την ηγεσία σας. Ε, τα αποτελέσματα ε, ήταν σημαντικά. Έχετε αφιερώσει πάρα πολύ ευφυΐα και πάρα πολύ χρόνο και πολύ δημιουργικότητα, γιατί πρέπει να είμαστε και δημιουργικοί βάσει των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και το κάνετε αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα ολόκαρδα να σας ευχαριστήσω γιατί με τις δράσεις σας ε, αναφερθήκατε άλλωστε και στο θετικό πρόγραμμα, ε, τις διάφορες, ε, τις διάφορες διαδικασίες. Πάντοτε χρησιμοποιήσατε το διάλογο για αμοιβαίο συμφέρον και εξασφαλίσατε να υπάρχει συνεχή δουλειά ανεξαρτήτων των προβλημάτων και των εμποδίων, να συνεχίζει λοιπόν συνεχώς η δουλειά. Ε, θα ήθελα να μας έλεγε ε, Ινσαλά ο κύριος Τσαβούσογλου όταν μας λέτε ότι το 2014 θέλουμε η έκθεση προόδου να είναι σημαντικότερη και καλύτερη από, το 2013, από το 2013. Ε, πραγματικά υπολογίζουμε πάρα πολύ σε εσά, βασιζόμαστε σε εσά για να προχωρήσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία. Θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες το απόγευμα σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις ε, για το δικαστικό τομέα. Δεν ξέρω εάν ο ε, πρέσβης θα ήθελε να προσθέσει κάτι εκ μέρους του ε, Συμβουλίου. Μια και ο Επίτροπος ανέφερε το ζήτημα αξιοπιστίας από αμφότερες τις πλευρές. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν σχολιάζω κράτη μονομένα, κράτη με μέλη και τις θέσεις τους. Δεν είναι αυτή η θέση μου και η προσέγγιση μου. Η τρέχουσα, αλλά φαντάζομαι και η προσεχή η Ιταλική Προεδρία με πολύ μεγάλη χαρά θα ανοίξει και άλλα κεφάλαια. Υπάρχουν κεφάλαια που δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν γιατί η Τουρκία μας λέει ότι δεν είναι έτοιμη να τα ανοίξει. Υπάρχουν άλλα κεφάλαια που δεν ανοίγουν γιατί το Συμβούλιο δεν θέλει να τα ανοίξει. Είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ότι μια εξέλιξη στην, ε, στο Κυπριακό θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα και το πιστεύω ακράδαντα. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν πιστεύω θα ανοίξουμε κεφάλαια στους επόμενους μήνες. Είμαστε όμως 28, όχι 27. Πιστεύω και αισιοδοξώ ότι στους προσεχείς μήνες θα ακούσουμε καλές ειδήσει και ότι θα ανοίξουν και άλλα κεφάλαια. Αυτή είναι και η τελική μου παρατήρηση. Η Πρόεδρος, αγαπητέ κύριε Πρέσβη, το, το ελπίζουμε όλοι, το ελπίζουμε όλοι και σας ευχαριστώ. Οι προσκεκλημένοι μας θα αποχωρήσουν. Τους ευχαριστώ για την παρουσία τους, για την ποιότητα, για το ευήκον, για την διαθεσιμότητα να απαντήσουν και προτείνω να τους ε, να τους χειροκροτήσουμε θερμά για να τους ευχαριστήσουμε. Uh, Ο κύριος Δεμίρκρον, θα ήθελα ιδιαιτέρως να πω στον κύριο Φίλε, μια και είναι κατά πάσα πιθανότητα η τελευταία μας κοινή συνεδρίαση, να... ένα θερμό ευχαριστώ γιατί δεν μας αφήσατε ποτέ μόνος μας. Με μεγάλη αποφασιστικότητα και στράτευση βρεθήκατε στο πλευρό μας. Ήσασταν συνοδοιπόρος, δώσατε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, ιδιαίτερα η τουρκική πλευρά και ως συμπρόεδρος εγώ προσωπικός θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Και θα ήθελα να πω ότι με πολύ μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα επεξεργαστήκατε όλες τις εκθέσεις που εκπονήσατε για την Τουρκία. Η προσοχή που αναμένετε το Μάιο θα είναι η τελευταία σας. Ελπίζουμε όπως και οι προηγούμενες και αυτή να είναι καλά, εξισορροπημένη, αντικειμενική, επικοδομητική, θετική και μια έκθεση η οποία θα επισημαίνει βεβαίως τις ελλείψεις. Σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα είναι τέτοια η έκθεση. Θα ήθελα επίσης ε, να ευχαριστήσω και τον Προεδρεύοντα ε, και μέσω αυτού και την ε, Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον Τούρκο πρέσβη που είναι παρόν και τον κύριο Υπουργό βεβαίω. Εκ μέρου τη Συμπροέδρου, νομίζω μπορώ να κηρύξω το πέρα αυτού του μέρου τη συνεδριάσεω, τουλάχιστον όσο να επιτρέψουμε στου προσκεκλημένου μα να αποχωρήσουν. Η κυρία Φλότρο, όχι, όχι, όχι, καθίστε, μην φεύγετε. Έχουμε να οργανώσουμε κάποια πράγματα. Μην φύγετε. Διακόπτω μόνο για να χαιρετήσω, να ε, αποχαιρετήσω τους προσκεκλημένους.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 Euh, chers collègues, on va reprendre les travaux pour organiser la suite de notre commission. Παρακαλώ να ξαναρχίσουμε για να οργανώσουμε και τις υπόλοιπες εργασίες της Επιτροπής μας. Μήπως μπορείτε να καθίσετε παρακαλώ. We come back at the session. Να ξαναρχίσουμε παρακαλώ να οργανώσουμε το τελευταίο τμήμα της ε, συζήτησής μας. Παρακαλώ καθίστε.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 Γκίζλι Γκιντέρ και η Σίκ, αν είναι εδώ, Ο, θέλετε να πάρετε το λόγο. Madame Inchekara, on entend que vous. Κυρία Ιντσέκαρα, μόνο εσείς ακούγεστε. Monsieur Ishik, est-ce que vous souhaitez toujours... Do you want to... Κύριε Ishik, θέλετε να πάρετε το λόγο? You still want to take the floor? Θέλετε να πάρετε το λόγο, κύριε Ισικ. Επαναλαμβάνω. You don't want to take the floor. Okay. So, uh, I have another... Ναι, θέλετε. Υπάρχει άλλος ένας συνάδελφος που θέλει να λάβει το λόγο. Ο κύριος Γκισλίγκιντερ. Όχι. Καλά. Ωραία. Τότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο τμήμα της συνεδρίασή μας ε, σε σχέση με τον πολιτικό διάλογο υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον, πολύ καλή η συζήτηση αυτή και χρήσιμη για, γιατί πολλά θέματα αποσαφηνίστηκαν και θα ήθελα τώρα να οργανώσουμε το τελευταίο τμήμα της συνεδρίασής μας Έχουμε ακόμη μια συζήτηση για τις ε, δικαστικές μεταρρυθμίσεις το απόγευμα. Δυστυχώ όμως δεν θα είναι παρόν ο Υπουργός ε, Δικαιοσύνης, όπως τώρα όλοι γνωρίζουμε. Έχουν επίση παρουσίαση της κατάστασης των διαπραγματεύσεων για το ε, κεφάλαιο που αφορά το περιβάλλον. Και αύριο το πρωί την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας και για την Τελωνιακή Ένωση. Αυτά. Θα θέλαμε, ο κύριος Δεμιρκυράν και εγώ, θα θέλαμε να, να οργανώσουμε σήμερα το απόγευμα όλες μας τις, συνεδριά, τις ε, ε, συζητήσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την οργάνωση. Όλοι οι εμπειρογνώμονες ε, μπορούν να είναι παρόντες. Βέβαια δεν θα είναι πολλοί ευρωβουλευτές παρόντες γιατί όπως γνωρίζετε ε, υπάρχει προεκλογική εκστρατεία αυτή τη στιγμή και πολλοί συνάδελφοι απουσιάζουν. Φοβάμαι λοιπόν ότι δεν θα είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι παρόντες. Ελπίζω να ολοκληρώσουμε όλες μας τις συζητήσεις σήμερα το απόγευμα και τα τρία θέματα που μας έχουν μείνει. Μπορούμε να αλλάξουμε κατά αυτόν τον τρόπο την ημερήσια διάταξη. Δεν δημιουργεί πρόβλημα αυτό για σας. So, um, I think we can begin with the reforms. Άρα μπορούμε να αρχίσουμε με τον εκδημοκρατισμό, τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις και το άνοιγμα του κεφαλαίου, των κεφαλαίων 23 και 24. Το καλύψαμε ήδη σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπούμε σε λεπτομέρειες και να περάσουμε στις ε, συμφωνίες, ε, ε, στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και στο, στην Τελωνιακή Ένωση στη συνέχεια και στο τέλος να περάσουμε στην κατάσταση των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 27, το περιβάλλον, τμήμα 1. Συμφωνείτε κι εσείς? Ωραία. προτείνω να Μισό λεπτό διορθώνει η Πρόεδρος ε, και διακόπτη ε, λέγοντας ε, ότι πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 73ης συνεδρίασής μας. Θα σας ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσεις, οπότε τα εγκρίνουμε ως έχουν, αν δεν έχετε παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε τώρα να κλείσουμε την πρωινή μας συνεδρία. Έχετε όλες τις πληροφορίες για το μεσημεριανό γεύμα. Ωραία. Τα λέμε εκεί τότε.